colleagues, I would like to start the meeting. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Because we are already late, so could we please start the meeting? Thank you very much indeed. Now we start... Ευχαριστώ πολύ και τώρα ξεκινάμε την τακτική συνεδρίαση που έχει να κάνει με τη συζήτηση για το Brexit. Έχουμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Καταρχάς ε, θα ακούσουμε τον Γκί Φέρχοφστατ που είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαδικασία του Brexit, μέλος της Επιτροπής ΑΦΚΟ και θα ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει ως τακτική ενημέρωση, γιατί πρόσφατα έχουν συμβεί πολλά. Και επίσης, όπως ξέρετε, αυτή η Επιτροπή έχει έναν πολύ σημαντικό ριζόντιο ρόλο στη διαδικασία. Στο τέλος της διαδικασίας η Επιτροπή θα κάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, των αποφάσεων και θα υπάρξει μια πρόταση στην Ολομέλεια να προσυπογραφούν τα αποτελέσματα. Θα αρχικούσουμε λοιπόν πρώτα τον Γκί Φέρχοφστατ και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις. Μετά θα ακούσουμε τον καθηγητή Πογιάρες Μαντούρο για τις επιπτώσεις και τις νομικές επιλογές ε, που ε, υπάρχουν ε, για τη διαδικασία του Brexit. Γκί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σου δίνω το λόγο. Ελπίζω μετά να έχουμε και πέντε λεπτά για τις, απαντήσεις, για τις ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεση της Επιτροπής. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση να σας δώσω μια νέα επισκόπηση του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Είναι το follow-up μιας προηγούμενης έκθεσης, μιας αναφοράς που έκανα πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, όταν προετοιμάσαμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τον Brexit. Μπορώ ίσως να ξεκινήσω θυμίζοντάς σας ότι αυτό το ψήφισμα που ετοίμασε η διάσκεψη των Προέδρων και υποστηρίχθηκε από πέντε πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία, 560 ψήφους, ε, υπέρ, 133 κατά και 50 αποχές. Νομίζω ότι δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι αυτό το ψήφισμα υπήρξε και η βάση για τις ε, διαβουλεύσεις και αργότερα για την εντολή που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το περασμένο Σάββατο. Η συνάντηση του Συμβουλίου για την εντολή διήρκησε τέσσερα λεπτά. Το γεγονός αυτό νομίζω αποτελεί σημάδι της καλής προετοιμασίας ε, που είχε γίνει για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, μέσω του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Όταν συγκρίνεται το ψήφισμα του Κοινοβουλίου με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια ομοιότητα. Όχι μόνο σε επίπεδο περιεχομένου, αλλά και στην ε, διατύπωση. οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ δηλαδή, ο κύριος Μπρόκ και ο κύριος ε, Κολτχέρη με την ε, βοήθεια των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, λάβαμε μέρος στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις για να οριστικοποιήσουμε το κείμενο που εγκρίθηκε στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Σάββατο. Δεν θα σας αναφέρω τώρα όλα τα στοιχεία του ψηφίσματος, ή το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών, το γνωρίζετε αυτό. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό σε επόμενη φάση είναι να αποφασίσουμε τι θα παρουσιάσει σήμερα ο κύριος Μπαρνιέ, ο διαπραγματευτής, μετά από την συνάντηση του Κολεγίου των Επιτρόπων ε, σχετικά με τις οδηγίες ε, για την διαπραγμάτευση είναι ένα non-paper, μια πρόταση που έχει τεθεί ήδη στη διάθεσή σας από την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν έλαβα εγώ το κείμενο ε, για αυτές τις ε, οδηγίες, το έστειλα αμέσω, το διαβίβασα στις διάφορες εμπλεκόμενες επιτροπές, διότι στην πραγματικότητα αυτές οι οδηγίες ε, έχουν να κάνουν με λίγα συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Ε, πρώτον, το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, με ό,τι αυτό ενέχει θα είναι το πρώτο μπλοκ των οδηγιών διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο μπλοκ έχει να κάνει με τον οικονομικό διακανονισμό και σχετικά με, με τις λεπτομέρειες αυτού θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Δεύτερον, ε, τρίτον, συγγνώμη, ε, κάποια θέματα σχετικά με την ε, συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη μελλοντική αποχώρηση και το κεφάλαιο για τις διοικητικές διαδικασίες. Και τέλος, η εποπτεία της όλης διαδικασίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά είναι τα πέντε στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτές τις ε, λεγόμενες οδηγίες διαπραγμάτευσης. Να σας ενημερώσω επίσης, αγαπητοί βουλευτές ε, της Επιτροπής ΑΦΚΟ, ότι θα παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Από την έγκριση του ψηφίσματος έχουμε θεσπίσει το Brexit Steering Group, τη διευθυντήρια ομάδα που έχει εκπροσώπους των πέντε πολιτικών ομάδων των πέντε ομάδων που στήριξαν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, βέβαια, όπως είναι φυσικό, υπάρχει και η δική σας παρουσία ως Πρόεδρο της ΑΦΚΟ, διότι η ΑΦΚΟ πρέπει να έχει την γενική επισκόπηση αυτής της διαδικασίας. Η παρουσία σας λοιπόν στο steering group είναι πάρα πολύ σημαντική για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, αυτό το σκόπο. Σήμερα η Επιτροπή θα παρουσιάσει λοιπόν μία πρόταση για αυτές τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που θα έχουν αυτά τα πέντε στοιχεία για τα δικαιώματα των πολιτών, τον, ε, διακανονισμό, τον οικονομικό διακανονισμό, για τα σύνορα και συγκεκριμένα τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, τις διοικητικέ διαδικασίες και την εποπτεία της διαδικασίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτή η πρόταση θα εγκριθεί στην συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 22 Μαΐου. Η διάσκεψη των Προέδρων προτίθεται επισήμως να αντιδράσει σε αυτή την πρόταση του Κολεγίου των Επιτρόπων στις 11 Μαΐου. Πριν δηλαδή τη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 22 Μαΐου. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι για, την, για το steering group που ασχολείται με το Brexit είμαστε σχεδόν 100% ευθυγραμμισμένοι με την πρόταση του non-paper που ο Μπαρνιέ θα παρουσιάσει σήμερα την ανεπίσημη πρόταση δηλαδή στο Κολέγιο των Επιτρόπων για τα διάφορα αυτά θέματα. Και για αυτό το λόγο ζητήσαμε από τις επιτροπές μας, τις ειδικέ επιτροπές, ε, τις αρμόδιες επιτροπές να λάβουν ε, αυτά, αυτό το non-paper ε, για ε, οι επιτροπές είναι η ΕΜΠΛΕ, η ΛΥΜΠΕ, η Γιούρι και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Πολιτών. Έχουμε στείλει το κεφάλαιο για τον οικονομικό διακανονισμό στην, στις δύο επιτροπές για τον προϋπολογισμό την Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και φυσικά Όλα αυτά τα κείμενα έχουν αποσταλεί και στην κυρία Χιμπνερ, την ε, πρόεδρο της δικής μας επιτροπής, ε, για να ε, δούμε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι αντιδράσεις από τους Προέδρους των Επιτροπών ήταν όλες θετικές, δεν υπήρχαν θεμελιώδεις παρατηρήσεις ή κριτικές επικρίσεις για το κείμενο του ανεπίσημου εγγράφου του non-paper που προτείνει ο κύριος Μπαρνιέ. Παρόλα αυτά εχθές στο steering group για το Brexit μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ κάναμε κάποιες πιο συγκεκριμένες και απτές προτάσεις που θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εάν χρειάζεται θα ε, διατυπωθούν και στις 11 Μαΐου από τη διάσκεψη των Προέδρων ως ε, επίσημη θέση αυτών για να τις έχει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 22 Μαΐου. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης που εμείς κάθε φορά επαναλαμβάνουμε είναι μια προσθήκη ε, σε αυτές τις οδηγίες διαπραγμάτευσης είναι το θέμα των συνόρων και της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά να ορίζουμε ότι αυτό αφορά σε όλα τα μέρη της συμφωνίας αυτής. Αυτό είναι κάτι που έχει προσθέσει το Κοινοβούλιο από την πρώτη μέρα και πρέπει να ληφθεί υπόψη και στις οδηγίε διαπραγμάτευση. Είναι ήδη στι κατευθυντήριε γραμμές όπως ξέρετε, αλλά να μπει και στις οδηγίε διαπραγμάτευση. Δεύτερον, για τα δικαιώματα των πολιτών, επίσης είπαμε ότι η εντολή ε, των Βρετανών ε, στα Συμβούλια των Εργαζομένων και στις Επιτροπές Εργαζομένων θα πρέπει να διατηρηθούν να μην υπάρχει πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας ε, το οποίο ε, έχει θεσπιστεί και έχει εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό ως προσθήκη στις οδηγίες Επίσης, ε, κάτι άλλο που ήταν σημαντικό είναι μια άλλη πρόταση του Κοινοβουλίου σε όλο το θέμα των ε, δικαιωμάτων των ε, πολιτών θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα εξ αρχής και έως το τέλος. Ως Κοινοβούλιο έχουμε συμφωνήσει και έχουμε επιμείνει στο να αποτελέσει το κεφάλαιο αυτό, το πρώτο κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να, με μια κατάσταση στην οποία εκατομμύρια Βρετανών και Ευρωπαίων πολιτών ζουν στην αβεβαιότητα όπως σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν και συμφωνήσαμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο ένα της διαπραγμάτευσης. Όμως είχαμε κάποιες προτάσεις ε, που ε, θέσαμε για να συμπληρώσουμε τις οδηγίες διαπραγμάτευσης σε αυτό το θέμα. Για το θέμα του οικονομικού διακανονισμού, φυσικά επαναλάβαμε τη θέση ότι που, που έχουμε ήδη υπογραμμίσει στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή να τηρηθούν οι δικές, όλες οι δεσμεύσεις, όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων, ακόμα και αυτές ε, που είναι πιο έκτακτες. Ε, με τέτοιο τρόπο, ώστε ο οικονομικός διακανονισμός και τα διάφορα ε, στοιχεία αυτού να προσεγγίζονται σωστά κατά τη διαπραγμάτευση. Για την εποπτεία της όλης διαδικασίας, το Κοινοβούλιο έχει προτείνει, βάσει, και στη δική, βάσει της δικής σας πρότασης, κυρία Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην όλη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα είναι αυτό που θα ε, δρά ως επόπτης Υπάρχει αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές ε, που εγκρίθηκαν το Σάββατο, θέλουμε να είναι και στις οδηγίες διαπραγμάτευσης. Και τέλος, Έχουμε προτείνει στην Επιτροπή και αν είναι απαραίτητο θα το επαναλάβουμε και στις 22 Μαΐου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ότι με την εισαγωγή των οδηγιών διαπραγμάτευσης καλό θα ήταν να εισαγάγουμε και μία αρχή. Ότι δηλαδή οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνονται καλή τυπίστη και δεν θα πρέπει να παρακολύεται η καθημερινή ε, λειτουργία και οι δραστηριότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό μπορεί να γίνει πρόβλημα, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα με τις διαμάχες σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά σταμάτησαν και τέθηκαν σε αναμονή ε, των αποφάσεων για τον Brexit. Ε, το έχουμε ήδη θέσει λοιπόν ε, στην Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα μπει στην πρόταση που θα εγκριθεί σήμερα από τους Επιτρόπους. Μια ξεκάθαρη αναφορά στην εισαγωγή αυτών των οδηγιών ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε η τακτική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τίθεται εν αμφιβόλο λόγω ε, αυτών των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Τώρα για την αλληλουχία των ε, διαπραγματεύσεων, κυρία Πρόεδρε, η πρόταση που έχουμε κάνει στο ψήφισμα μπήκε στις κατευθυντήριες γραμμές και θα επαναληφθεί και στις οδηγίες διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φάση έχει να κάνει με τη συμφωνία αποχώρησης και όταν θα έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος στην πρώτη αυτή φάση και μόνο τότε θα μπορούμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε τη δεύτερη φάση, τη μελλοντική σχέση δηλαδή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και η ΑΦΚΟ νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Διάσκεψη των Προέδρων με την πρότασή τους προτίθενται να έχουν μια δική τους αξιολόγηση στο δεύτερο μισό του έτου σχετικά με την επαρκή πρόοδο. Αν υπάρχει δηλαδή και μπορούμε να πάμε από τη φάση 1 στη, στη φάση 2. Στην πραγματικότητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι που θα πρέπει να λάβει αυτή την απόφαση γιατί αυτοί αποφασίζουν για τις κατευθυντήριες γραμμές. Όμως θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο έχει ως ρόλο και ως ευθύνη να γνωμοδοτήσει ε, εν ευθέτω χρόνο για το αν έχει υπάρξει υπαρκής πρόοδος. Αυτό μπορεί να είναι τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Δηλαδή, πέραν του ψηφίσματος που εγκρίναμε πριν από μερικές εβδομάδες, καλό θα ήταν να έχουμε και ένα δεύτερο, όπως το αποκαλώ, οριζόντιο ψήφισμα σχετικά με το εάν έχουν, έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος για να μπορέσουμε να πάμε από τη φάση 1 στη φάση 2 των διαπραγματεύσεων και αυτό το ψήφισμα να εγκριθεί πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταθέσει τη δική του αξιολόγηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξουμε. Να δούμε εάν εντός των κατευθυντηρίων γραμμών και των οδηγιών διαπραγμάτευσης μπορούμε να έχουμε την επαρκή πρόοδο που θα μας πάει από τη φάση 1 στη φάση 2 η οποία θα σημάνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το δεύτερο αυτό θέμα, το τελευταίο αυτό θέμα, να σας θυμίσω συνάδελφοι, ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του από την πρώτη κιόλας μέρα έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή. Ε, μιλήσαμε ε, για το άρθρο 217 της Συμφωνίας Σύνδεσης ως ε, το άρθρο πλαίσιο, γιατί είναι ευέλικτο, μπορεί κανείς να κάνει πολλά μέσα στα πλαίσια μιας ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι μικρή, ευρία, μπορεί να είναι μόνο για το εμπόριο και την οικονομία, αλλά μπορεί να είναι και για την ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική. Από τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και μετά έχουμε ένα πλαίσιο που μας δίνει πολλά πράγματα, πράγματα που δεν είχαμε στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένα όμο ξεκάθαρο πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ως συμβουλή στην ΑΦΚΟ, στο Steering Group ε, για, την, ε, για το Brexit, στη διάσκεψη των Προέδρων, σε όλα τα άφορα. συμφωνούμε και λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε βάσει αυτής της γραμμής. Η συμφωνία σύνδεση δηλαδή να θεωρείται ως το κατάλληλο πλαίσιο για αυτή τη μελλοντική σχέση με το Ενωμένο Βασίλειο. Έτσι λοιπόν, το επόμενο βήμα για μας είναι φυσικά η προετοιμασία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με δική σας ε, παρουσία στο Brexit Steering Group. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Φυσικά θα σας παρακαλέσω να, είσαι, να είστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί και σύντομοι στις παρεμβάσεις. Ο γκεωργ Σέφλινγκ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φερχόφστατ ε, για το έργο του και για την παρουσία του εδώ σήμερα. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η παρουσίαση της κατάστασης ε, ως έχει μέχρι στιγμής. Ε, καταρχάς θα ήθελα να κάνω δύο γενικές υποδείξεις. Η πρώτη είναι ότι η μη διαπραγμάτευση ε, Μάλλον η διαπραγμάτευση υποτίθεται ότι καταλήγει εκεί που θέλουν να την πάνε οι διαπραγματευτές. Υπάρχουν βέβαια και κάποια πρόβλεπτα, οι αστάθμητοι παράγοντε, όπω είναι η προκήρυξη εκλογών από την κυρία Μέη. Το θέμα είναι ε, πώ θα ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία. Τι θεωρεί ο κύριο Φερχόφ αυτά, αυτά τα πέντε σημεία τα οποία ανέφερε. Πολύ σωστά δε. Ε, πώς θα περάσουν αυτά τα πέντε σημεία ε, τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεύτερον, πόσο θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο το ρόλο του Κοινοβουλίου για τα θέματα που έχουν σημασία, διότι έχω την εντύπωση ότι δεν το έχουν αντιληφθεί πλήρως, ελπίζω να κάνω λάθος. Και τρίτον, αυτό που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και το 5 για το ρόλο του δικαστηρίου. Τον του Ευρωπαϊκού. Φαντάζομαι ότι αυτό που θέλουμε είναι από νωρί να, διαπραγμα... να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία το δικαστήριο, αλλά δεν το θέλουν οι Βρετανοί. Φαντάζομαι ότι εκεί θα έχουμε σύγκρουση. Ε, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο κύριος Φερχόφστατ και ένα ερώτημα που μπορεί και να μην απαντήσετε αν δεν θέλετε, αλλά αν είχατε τη μηχανή του χρόνου. Το άρθρο 50 πώς θα το είχατε συντάξει, όπως ε, είναι τώρα, τελείως διαφορετικό, θα ήταν ε, ριζικά διαφορετικό. Έχω και εγώ την εμπειρία μου ε, και τις απόψεις μου. Εσείς θεωρείτε ότι το άρθρο 50 στην παρούσα του μορφή είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάκελ Μπόνι τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φερχόστατ για την παρουσίαση και το έργο του μέχρι τώρα. Δεν έχω πολιτικά σχόλια, αλλά θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχέση με τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να δούμε και το διατομεακό έργο για κάποια ζητήματα, όπως ε, παραδείγματος χάρτη δικαιωμάτων των πολιτών. Διότι αναζητούμε ίσως κάποιες λύσεις πολύ πιο πολύπλοκες, όπως είναι η προστασία της ιδιωτικότητας, τα μελιώδη δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το εμπόριο, για την άπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τον κανόνα της αμοιβαιότητας ε, για τους πολίτες, ένθεν κακήθεν και για την υπηρετική Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε να εφαρμόσουμε και τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, έχουμε τον κανονισμό για την ιδιωτικότητα που επεξεργαζόμαστε. Πώς θα δημιουργήσουμε ένα είδος ε, διατομεακής, δια, διεπιτροπιακής, αν μπορώ να την πω, συνεργασίας για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζέιμς. Uh, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φερχόφστατ που ήρθε σήμερα το πρωί Κύριε τα άκουσα αυτά που είπατε ε, και ακολουθείτε σκληρή γραμμή και θέλω να το στηρίσω, να το συγκρίνω αυτό που λέει ο αρχηγός των Lib ε, Dem στην, ε, στη Βρετανία. Δεν ξέρω μήπως πήρατε από αυτόν παράδειγμα και μερικά από αυτά που είπατε, είχατε επαφή μαζί του. Τέλος πάντων, αυτό που ανησυχεί πολλούς που ήρθαν σε επαφή μαζί μου ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να κάνει με το ότι αναγνωρίζουν ότι εδώ έχουμε μια διαπραγμάτευση και οι δύο πλευρές αναφέρουν ποιες είναι οι παράμετροι, ποιες είναι οι θέσεις τους, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τους και αυτό είναι φυσιολογικό, δεν έχουμε πρόβλημα ως προς αυτό το πλαίσιο. Όμως αυτό που νομίζω ότι έχει οξύνει τα πράγματα ε, και δημιουργεί ένταση στην κοινή γνώμη είναι τι έγινε μετά τη συνάντηση Γιούνκερ και Βρετανίδας Πρωθυπουργού και το ότι διέρευσαν στον τύπο, από ό,τι φαίνεται κάποια σχόλια, και υπάρχει ένα συνεχής εκφοβισμός ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, λένε, ε, βγήκαν όλα αυτά τα σχόλια προς τα έξω. Εγώ θα ήθελα να τα σχολιάσω τα λεφτά στηρίζετε αυτή τη θέση που βγήκε προς τα έξω το Σαββατοκύριακο ή στη δική σας θέση, εφόσον είστε κανείς από τους βασικούς διαπραγματευτές, θα παρακαλέσετε να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ηρεμία, να χαμηλώσουν οι τόνοι γιατί νομίζω ότι αυτό που ίσχυε μέχρι το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το φιλικό διαζύγιο κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ρωτώ τον κύριο Φερχόφστατ αν έχει την εντύπωση σε σχέση και με αυτά που είπε ο κ. Σέρτφλιν, να καταλαβαίνουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βρετανία. Καταλαβαίνουν γενικά τη διαδικασία, αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Γιατί ενίοτε μας δημιουργείται εντύπωση ότι έχουν μια εντελώ διαφορετική διαδικασία διαπραγμάτευση στο μυαλό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καταθέσει επιτάπτως. Και δεύτερον, η Βρετανική κοινή γνώμη ε, διακατέχεται από ευτυχή άγνοια ακόμη για το τι ε, απαιτείται σε διάφορα μέτωπα για αυτές τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή ε, τελικά τι θα ζητήσει ε, η Βρετανική κυβέρνηση. Θα ζητήσει να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση κάποιες πτυχές τουλάχιστον. Προτίθεται να ζητήσει κάποιο είδους συνέχιση στη συμμετοχή στις ε, παρουσιάσεις των οργανισμών για την αεροπορία, τον Οργανισμό φαρμάκων, σε εκτελεστικούς οργανισμούς τέλος πάντων. Ναι ή όχι. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι μεταβατικέ διευθετήσει, παραδείγματο χάρη για τον τομέα της Αλίας ή τη γεωργίας. Πολλά ακόμη δεν έχουν ξεκαθαριστεί από τη Βρετανική κυβέρνηση. Ούτε καν στο κοινοβούλιο της χώρας και στους πολίτες της χώρας δεν είναι σαφή αυτά. Τι ενδείξεις έχετε, αν έχετε, ε, για τις προθέσεις ε, της Βρετανικής πλευράς. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Ο Γιώλα είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Γκί Φερχόφστατ για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω ότι ο Γκί μας εκπροσωπεί με πάρα πολύ ικανό τρόπο παρά τις επιθέσεις του UKIP που δεν θα πρέπει να μας πτωίσουν και να μας ανησυχήσουν. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Από το γεύμα Γιούν και βγήκε και είπε ότι έχω την εντύπωση ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι σε έναν άλλο γαλαξία, όχι σε πλανήτη άλλο δηλαδή βρίσκονται, αλλά και σε άλλο γαλαξία. Είναι δηλαδή έτη φωτός μακριά από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ. Το ρώτησε ε, και ο συνάδελφος ε, Ρίτσαρτ, ε, νομίζω ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει, σε ποιο γαλαξία βρίσκονται οι Βρετάνοι διαπραγματευτέ σε σχέση με μας. Και εδώ έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι στη συνθήκη έχουμε το άρθρο 217 που λέει ότι οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να ε, έχει καθεστώς συνδεδεμένης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εφόσον μια χώρα θελήσει τέτοιο καθεστώς, μπορεί να είναι μια χώρα ε. δεν μας βοηθάει το άρθρο αυτό. Και με αυτό το άρθρο ανησυχώ λίγο μήπως προβούμε σε μια διαδικασία σταχυολόγησης. Μπορεί να αρέσουν 10 σημεία, που και 20 να μην τους αρέσουν και έπειτα διαπραγματευόμαστε μία ε, συμφωνία με βάση το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι μια από τις κατευθυντήριες γραμμές ήταν ότι η χώρα που αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση από τις χώρες μέλη της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε μήπως συνεχιστεί αυτή η σταχυολόγηση. Το είδαμε άλλωστε και μέχρι τώρα να το κάνουν οι Βρετανοί και δεν θέλω να συνεχιστεί. Δεύτερο, τρίτο θέμα μάλλον, διαφάνεια. Από το γεύμα στην Downing Street έμαθα ότι η Βρετανική πλευρά θα ήθελε να μην είναι φανερά τα έγγραφα τοποθέτηση στα διάφορα position papers, αντίθετη είναι η ε, δική μας άποψη, όπως και με τις διαπραγματεύσεις ή τα TTIP. Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Θα ήταν γελίο να είναι μυστικές οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αντιθέτως πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο ανοιχτές, πιο διαφανείς. I would like to speak Polish. Um, θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ. Μια πολύ απλή σύσταση είναι να είμαστε πιο ορθολογικοί και να χαμηλώσουμε τους τόνους, γιατί πράγματι αυτό θα βελτιώσει το κλίμα των διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά και έχει κάθε δικαίωμα να διαδραματίσει το δικό του ρόλο στην όλη διαδικασία. Ωστόσο, το καλύτερο θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρήσει και αυτό ότι συμμετέχει, έχει ευθύνη στην όλη διαδικασία και για το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω είναι προς ε, το καλύτερο όφελος και προς το συμφέρον της Ευρώπης συνολικά να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία βάσει αμοιβαία ε, συνεννόησης. Φυσικά και δεν πρόκειται να βγουν όλοι κερδισμένοι και οι δύο πλευρές. Το θέμα είναι αν μπορούμε να ελεξιτοποιήσουμε, αν μπορώ να το θέσω έτσι, τις παράπλευρες απώλειες. Τα αρνητικά σχόλια που κατέστρεψαν την ατμόσφαιρα δυστυχώς διατυπώθηκαν και από τις δύο πλευρές. Και το πρώτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αμέσως μετά το δημοψήφισμα, για να δώσω ένα παράδειγμα, επίσης περιλάμβανε κάποια σχόλια ε, που ήταν φορτισμένα και σίγουρα δημιούργησαν αγανάκτηση και δεν βοήθησαν ε, στην εμπέδωση ενός καλού κλίματος. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε λοιπόν ευθύνη για το πώς θα διεξαχθεί όλη η διαδικασία και η εκτιμήση του κ. Φερχόφστατς ό,τι αφορά τη διαδικασία και συγκεκριμένα η εκτίμηση του κ. Φερχόφστατ για την πρώτη φάση της διαδικασίας για το φθινόπωρο μιλάω, θα είναι σίγουρα μια αξιολόγηση πρακτική και δεν θα είναι να σμοχλώ άσκηση πίεση στον κύριο Μπανί και στους άλλους. Αυτό που χρειάζεται, παραλαμβάνω, είναι ηρεμία, κοινό νους, για να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική έκβαση για την Ευρώπη. Θετική έκβαση. δεν μπορούμε να ε, έχουμε την άποψη να λέμε στους Βρετανούς ότι ζουν σε άλλο γαλαξία ή να τους κρατάμε κακία τέλος πάντων. Κύριε Σπινέλη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ Γκίφερ Χόφστερ για την εξαίρετη σου εισήγηση. Και εγώ είμαι ικανοποιημένη, όπως και εκείνος, από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έπαιξε αυτό το ρόλο του επιταχυντή όσον αφορά τις θέσεις του Συμβουλίου. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για τα όσα είπε για το ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ακόμα και για μια ενδεχόμενη μεταβατική συμφωνία. Η ερώτηση που έχω να κάνω αφορά την θέση του Συμβουλίου που είναι λιγότερο ξεκάθαρη από αυτή του Κοινοβουλίου και να προτείνουμε έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών που δεν είναι το δικαστήριο. Μάλλον προτείνει το Συμβούλιο. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το κλίμα που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις και αυτές οι διάφορες διαρροές και αδιακρισίες. Ε, που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες και δεν με ανησυχούν οι επιθέσεις του UKIP. Με ανησυχεί αυτό που θεωρώ πως είναι μία θέση σκληρού Brexit από πλευράς όλων των μερών, δηλαδή και της Βρετανικής κυβέρνησης αλλά και της Ένωσης, της Ευρώπης δηλαδή των 27. Υπάρχουν προφανείς διαφορές όχι μόνο για τα δημοσιονομικά θέματα, αλλά και σε σχέση με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τούμπαλιν και όσο, καθώς και όσον αφορά την σταδιακή διαπραγμάτευση. Δηλαδή σε διαδοχικές φάσεις. Και αυτό με κάνει να φοβάμαι τα εξής και θέλω να ξέρω τι πιστεύει ο Γκί με κάνει να φοβάμαι ότι τα δικαιώματα δεν θα είναι εγγυημένα συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες όπως θα θέλαμε. Δεύτερον, τι θα γίνει, ε, ότι θα γίνουν ε, αντικείμενο παζαρέματος ε, για διάφορα άλλα τα δικαιώματα και εφόσον μπαίνουμε σε μια φάση σκληρού Brexit ότι δεν θα υπάρχει βούληση για να φτάσουμε σε μια συνετική συμφωνία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να επικρατήσει η αρχή ότι πρώτα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία για την αποχώρηση και μετά θα μιλήσουμε για τις μελλοντικέ σχέσεις. Όμως το ίδιο το άρθρο 50 Και εγώ πιστεύω πως κάποια μέρα θα χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε την χρονομηχανή και να το ξαναγράψουμε. Όμως το άρθρο 50 λέει επίσης πως οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τι θα κάνουμε στο μέλλον ενώ διαπραγματευόμαστε την έξοδο. Τελευταίο ερώτημα τώρα που συνδέεται με αυτό είναι θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύει ο Γκίφερ Χόφστερ για αυτή τη φράση που σε μένα φαίνεται πραγματικά παράξενη και που φαίνεται στις, εμφανίζεται μάλλον σε αποφάσεις του Συμβουλίου στις κατευθυντήριες γραμμές. Τίποτα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συμφωνία μέχρι ότου να έχουν συμφωνηθεί όλα. Nothing must be agreed until all is agreed. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η καλή βάση για τις διαπραγματεύσει, αλλά πραγματικά θα ήθελα να το καταλάβω με αυτό, γιατί είναι κάτι το που ήδη απορρίφθηκε στις διαπραγματεύσεις στην Νότια γιατί είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Κινδυνεύει κανείς να φτάσει σε τέλειο αδιέξοδο, αν ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχουμε και πέντε λεφτά για τις απαντήσεις και έχω ακόμα μιλητές. Πέδρο Σίλβα Περέιρα. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ολόψυχα τον ε, Γκίφερ Χώστατη για την εισήγησή του. Εγώ έχω σύντομες, αλλά, ένα σύντομο αλλά σημαντικό θέμα να θίξω όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και να αποσαφηνίσουμε κάτι. Κατευθύνες γραμμές που υιοθέτησε το Συμβούλιο που εργάζεται επί τη βάση του δικού μας ψηφίσματο, λέει ότι βεβαίω ε, την ημέρα της εξόδου ε, θα εφαρμοστεί η συνθήκη ε, για τα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά λέει επίσης ότι όσον αφορά τη μεταβατική ρύθμιση, λέει ότι αν ε, ληφθεί υπόψη μία περιορισμένη χρονική διάρκεια ε, εφαρμογή του κεκτημένου, θα χρειαστεί από την πλευρά της, ε, της Ένωσης να, μάλλον θα χρειαστεί να εφαρμόζονται όλα τα δικαστικά, δημοσιονομικά και όλα τα της Ένωσης. Αυτό σημαίνει και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, δηλαδή εφόσον αυτό το ακεί, το κεκτημένο ε, θα, θα διατηρηθεί και θα παραταθεί για τη μεταβατική περίοδο, τότε αυτό σημαίνει ότι και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να διατηρηθεί για τη ε, διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Ευχαριστώ η Mercedes ε, Μπρέσο. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ τον Κίφερ Χόφστατ για την σαφή και ξεκάθαρή του ε, εισήγηση. Έχω μια-δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την δημοσιονομική ρύθμιση. Έχουμε στη διάθεσή μας ε, ξεκάθαρες προτάσεις, ε, για, μάλλον διαπραγματευτικές θέσεις, προτάσεις για αυτά που συζητώνται, γιατί αυτό είναι ένα από τα καυτά ζητήματα. Και αν καταλαβαίνω καλά, ε, προκαλεί μεγάλες ε, συγκρούσεις σε αυτή την πρώτη φάση διαπραγματεύση. Επίσης ε, και εμένα με ανησυχεί το κλίμα που επικρατεί και κυρίως έχω την εντύπωση ότι αυτός ο γόρδιος δεσμός των δικαιωμάτων των πολιτών θα είναι πολύ δύσκολο να λυθεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Από αυτή την άποψη κάποια στοιχεία ε, που αφορούν την διαπραγματευτική θέση για τη δεύτερη φάση, για το πλαίσιο, πιστεύω πως είναι απαραίτητο να δοθούν και από πλευρά της Ένωσης, διότι... να μπορούν ε, οι πολίτες ε, να έχουν εγγυήσει για το τι συμβαίνει και τι θα ισχύει εδώ, για τον κοινόφνητο είναι δύσκολο να βάλει ένα σύνορο για το τι δικαιώματα θα έχει σήμερα και τι δικαιώματα θα έχει στο μέλλον. Και είναι κάτι πολύ δύσκολο να το καταπιεί η κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνουμε για το μέλλον, γιατί ευπλαίσιο θα δεχτούμε, ένα πλαίσιο όπου δεν θα τα κλείσουμε όλα και θα πάμε σε σχέσεις τύπου ΠΟΕ. Έτσι, όλοι οι Ευρωπαίοι συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών που διερωτώνται ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης όσον αφορά τους πολίτες θα ξέρουν καλύτερα τι να περιμένουν. Διαφορετικά πιστεύω πως είναι καλύτερο όταν θα οριστούν οι συμφωνίες να μπορέσουμε έτσι να διαπραγματευτούμε ε, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ήδη να ξεκινήσει να βάζει κάποια στοιχεία διαπραγματευτικά Σε Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντερσον και ο Φάμπιο Χέλμουτ Σόλτς. Παρακαλώ σύντομα συνάδελφοι, γιατί δεν θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα, σύντομα. Εμένα με ανησυχούν αυτές οι διαπραγματεύσεις Η κυρία Μέη λέει ότι μη συμφωνία είναι καλύτερη από κακή συμφωνία. Αλλά η Τερέζα Μέη ε, κάνει λάθος. Εάν δεν βρεθεί συμφωνία, αυτό θα είναι φρικτό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα είναι ε, Brexit τύπου μετοπικής. Ε, και θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εσείς κύριε Φερχώστα, ποιος είναι ο κίνδυνος για με τοπικού τύπου ε, σύγκρουσης Brexit. Ευχαριστώ. Ο Φάμπιο. Ναι, θα προσπαθήσω ε, θα να, είμαι, να είμαι λακωνικός. Πρώτη παρατήρηση να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την εισήγηση και με χαροποίησε το γεγονός ότι τα δικαιώματα των πολιτών μπήκαν στην πρώτη θέση Μόνο Ιταλίες, οι ε, Ιταλοί είναι πάνω από 300.000 στο περιοχή του ευρύτερου Λονδίνου ε, και φαντάζομαι και θα είναι και πολύ περισσότεροι ε, σε ολόκληρη τη χώρα. Ε, γι' αυτό και με χαροποιεί σας λέω το γεγονό ότι μπήκε πρώτο το θέμα αυτό και ότι δεν θα, δεν θα, αποτελέσει έτσι, δεν θα πέσει μάλλον θύμα παζαρέματος στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Έπειτα, όταν είπατε ότι ανάμεσα στο steering group, μάλλον ότι στο steering group συμφωνεί σχεδόν 100% με την πρόταση του Μπαρνιέ, ποια είναι η ενδεχόμενη διαφορά απόψεων σε σχέση με τη διαπραγματευτική θέση του εγγράφου του Μπαρνιέ. Δεύτερη μου ερώτηση, εάν δούμε εν μέρη το προβληματισμό της Μπάρμπαρα που συμμερίζομαι για το κινδύνο σκληρού Brexit, για τον κίνδυνο μάλλον σκληρού Brexit, θα ήθελα να ξέρω πόσο υπό το φως αυτών των φημών που όλοι διαβάσαμε στις εφημερίδες σήμερα Πόσο θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος ε, να υπάρξει σκληρό Brexit μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Και έπειτα, σε κάθε περίπτωση οι διαπραγματεύσεις φαίνεται πως θα είναι δύσκολες και σκληρές δεδομένες της απόστασης απόψεων ανάμεσα στα δύο μέρη. Πρακτικά έχετε όμως σκεφτεί πώς θα λύσετε το θέμα των μελλοντικών εκλογών όταν αυτές ε, θα γίνουν ε, και αυτή η παράταση των διαπραγματεύσεων δύο ετών ε, διαπραγματεύσεις που κανονικά θα έπρεπε να φτάσουν ε, στην έξοδο της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου συν μια προεκλογική διαδικασία για το, εξατία μάλλον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μόλις θα έχει κλείσει το Brexit. Ε, θα δούμε το μέλλον της Γεωργίας. Και επίσης αναφέρθηκε η αρχή της καλής πίστης Ότι δηλαδή η Βρετανία δεν μπορεί να κάνει διμερείς διαπραγματεύσει ούτε εμπορικέ ούτε αλλού τύπου, εφόσον αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουν συμφωνίες, ε, όμως εκείνοι ίσως ε, να το κάνουν με μια ρήτρα ανάκληση ε, στη φάση εφαρμογής δηλαδή αυτής της συμφωνίας να κάνουν τέτοιες δημορίες, αλλά επειδή έχει ενεργοποιηθεί το, το άρθρο 50 Δηλαδή, να, πω, να λένε οι Βρετανοί, αυτή η συμφωνία θα είναι έγκυρη μόνο όταν και αν βγούμε από την Ένωση. Μια τέτοια ρήτρα μπορεί να υπάρχει ή είναι σε αντίθεση με τη ρήτρα της καλής πίστης από νομική άποψη. Ευχαριστώ. Τελευταίο μονόλεπτο σχόλιο παρακαλώ από το Χέλμο του Σούλτσε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκί για την εισήγηση που μας έκανες. Νομίζω ότι είναι σαφές ε, με τις κατευθύνσεις γραμμές στο που βρισκόμαστε, αλλά μια ερώτηση για όλους μας και μάλλον για σένα, όλους ιδιαίτερους. Πώς, πώς είμαστε βέβαιοι ότι όλα, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι ότου όλα να συμφωνηθούν. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών δεν θα χρησιμεύσουν ως αντίβαρο για ε, υποχωρήσεις ή εκχωρήσεις σε άλλα κεφάλαια. Πώς είμαστε βέβαιοι ότι θα κρατήσουμε αυτή την πορεία. Δεύτερον, από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου επιφόσον είμαστε και έχουμε ήδη συζητήσει και με την ΕΠΑ για την ε, κοινότητα των ανατολικών αφρικανικών χωρών και των δυτικών αφρικών χωρών. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι θα σημάνει ε, το Brexit ε, για το μέλλον. Στην πράξη σε συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ε, ε, ε, δούμε πώς θα συζητήσουμε αυτές τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες αυτή τη στιγμή. Αυτές οι διαπραγματεύσεις επηρεάζουν και τις εμπορικές μας σχέσεις και για το μέλλον το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε και πάλι για το, με το στοιχείο για τον κίνδυνο ενός σκληρού Brexit. Συμφωνώ με τα σχόλια που έγιναν ότι θα είναι κακό για την Ευρώπη και θα είναι ακόμα χειρότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με στόχο να βρούμε μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα βασίζεται φυσικά στην ε, αρχή ότι ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορείς να είσαι σε καλύτερη θέση από ότι εντός. Αυτό το είπε και ο Τζο Λάινεν. Όμως, ε, ούτως ή άλλως, ένα άσχημο Brexit θα είναι κακό για όλους, κυρίως όμως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω. Το κλίμα δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, στη ζωή μου έχω κάνει διάφορες διαπραγματεύσεις. Όταν είσαι μερικές δεκαετίες στην πολιτική, έχεις κάνει διαπραγματεύσεις και στη χώρα μου. Και δεν με εκπλήσει αυτό που συμβαίνει τώρα. Πάντοτε γίνεται κάτι τέτοιο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Έτσι κλιμακώνεται η πίεση και από τις δύο πλευρές, για να είμαστε ειλικρινεί. Δεν θα αλλάξει αυτό μέχρι την 9η Ιουνίου, την ημέρα που πραγματικά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Άρα δεν με ανησυχεί τόσο αυτό, από, για την κλιμάκωση δηλαδή της πίεσης από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ευρώπης. Για μένα είναι δύσκολο να σας κάνω σχόλια σχετικά με το τι συνέβη στη συνάντηση μεταξύ Γιούνκερ και Μέη, γιατί δεν ήμουν εκεί. Αν δεν είσαι παρόν, δεν μπορείς να πεις κάτι για το τι συνέβη πραγματικά. Στα δικά μου μάτια, λοιπόν, ε, όταν έχουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις ε, έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα και αυτή η κλιμάκωση της πίεσης είναι κάτι που έχω δει δεκάδες φορές. Η δική μου ανησυχία είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που είπε και ο κύριος Κόρμπετ δηλαδή. Ποιες θα είναι τώρα οι προτάσεις από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δύσκολο να το αξιολογήσουμε αυτό προς το παρόν. Και αυτό μας ε, δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα δεν είναι καλή. Πάνω απ' όλα για τους πολίτες, γιατί για αυτούς είμαστε εδώ. Εδώ και ένα χρόνο οι άνθρωποι αυτοί είναι αβέβαιοι σχετικά με τα δικαιώματά τους, την κατάστασή τους, το καθεστώς που τους διέπει Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Το Κοινοβούλιο, όλοι μας έχουμε λάβει χιλιάδες email από ανθρώπους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Ευρώπη και ρωτούν τι θα συμβεί, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε λιγάκι. Πρέπει όσο μπορούμε να άρουμε αυτή την αβεβαιότητα ε, πριν ξεκινήσει ε, γενικότερα η διαπραγμάτευση να γίνει η έναρξη των διαπραγματεύσεων με αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στην συμφωνία για την αποχώρηση συνολικά. Γιατί όταν έχει συμφωνήσει για ένα πράγμα, στην ουσία φαίνεται ότι θα συμφωνήσεις και για το σύνολο. Στην πολιτική ε, σε αυτή την αρχή βασιζόμαστε συνήθως. Αυτό με ανησυχεί εμένα όμως. Δεν μπορούμε να ε, επιτρέψουμε να συνεχίσει αυτή η αβεβαιότητα για τους πολίτες μας μετά από ένα χρόνο, έξι μήνες. Διότι καταστρέφει ζωές, οικογένειες, επιχειρήσεις, το κοινοβούλιο πρέπει να μπει στην εμπροστοφυλακή για να το αποφύγουμε αυτό. Και αυτό κάνουμε τώρα στις οδηγίες της διαπραγμάτευσης. Ξεκαθαρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφάνεια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως ήδη έχει δημοσιευθεί το έγγραφο, ξεκαθαρίζει λοιπόν το πώς θα άρει αυτή την αβεβαιότητα για τους πολίτες. Ξεκινώντας ε, ε, με τους εργαζόμενους, τους αυτοπασχολούμενους, ε, τις οικογένειες, ε, μιλάμε για τα δικαιώματα διαμονής, κοινωνικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, κινητικότητας, αυτοπασχόλησης, αναγνώριση των διπλωμάτων, των πτυχίων, επίσημων τυπικών προσόντων. Ε, όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταδείξει έτσι με έναν ευρύ τρόπο, όχι στενό, ε, πώς θα, ε, πώς θα βλέπει, πώς θέλει να διαμορφωθούν. Και για να απαντήσω στην παρατήρηση του κυρίου Περέρα, για τον έναν ή τον άλλο λόγο υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Για παράδειγμα, ε, μια σταδιακή αποχώρηση από το κεκτημένο. Το κεκτημένο ε, διαρκεί για μια περιορισμένη περίοδο, maximum τρία χρόνια. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, αν συνεχίσουμε την ενιαία αγορά για αυτό το διάστημα, μιλάμε για όλη την ενιαία αγορά και την ελεύθερη κίνηση των ατόμων. Στη μεταβατική περίοδο δεν λέμε είναι μόνο για τα αγαθά αλλά όχι για τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος της διατύπωσης που αναφέρατε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Όλα τα βασικά στοιχεία του κεκτημένου συνεχίζουν. Και η ευαπτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι ε, συνεχίζει να υφίσταται και να ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί σήμερα και είναι σημαντικό από την πλευρά της Ευρώπης με πλήρη διαφάνεια να το δημοσιεύσουμε, γιατί έχουμε δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές, όλοι τις γνωρίζουν. Και μετά από την έκδοση, ε, από την έγκριση από το ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα δημοσιεύσουμε και τις οδηγίες διαπραγμάτευσης. Όλοι θα μπορούν να δουν, να αισθανθούν, να διαβάσουν ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα υπάρχουν μυστικές εντολές που θα έχουν δοθεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ε, στα τέσσερα θεσμικά όργανα γιατί αυτή η διαφάνεια είναι σημαντική. Είναι το κλειδί και είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά της Ευρώπης να την διατηρήσουμε. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τον χρηματοοικονομικό διακανονισμό. Κάποιοι λένε ότι είναι μια τιμωρία. Δεν είναι καμία τιμωρία η εκδίκηση. Απλώς όταν παίρνεις διαζύγιο δεν φεύγεις λέγοντας «Α, όλα τα βάρη στον σύζυγο, στον πρώην σύζυγο ε, και bye bye». Ε, δεν έχω χωρίσει ποτέ, δεν σας το λέω εξιδίας πείρας, αλλά κύριε Γκονζάλες Πόντς μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτά που λέω. Πρέπει να υπάρξει ένας οικονομικός διακανονισμός. Είναι προφανές. Και εμείς στο Κοινοβούλιο έτσι το βλέπουμε. Δεν έχουμε μπει σε καμία συζήτηση για κάποιο νούμερο. Εντάξει, υπάρχει εκεί για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα φανταστικό νούμερο. αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιες λογιστικές αρχές. Και αυτό είναι και στην πρόταση των ε, οδηγιών διαπραγμάτευσης, δηλαδή αυτές οι λογιστικές αρχές που θα αποτελέσουν τη βάση για τον διακανονισμό. Αν συμφωνήσουμε σε αυτές, τότε το νούμερο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των υπολογισμών. Ακόμα και αν είναι μη ρεαλιστικό. Ξέρετε πώς πάνε οι πολιτικές διαπραγματεύσεις. Και ο λόγος που πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτό δεν έχει να κάνει με την εκδίκηση ή την τιμωρία, έχει να κάνει με την ε, δικαιοσύνη, την τιμιότητα. Δεν μπορεί κανείς ε, να ζητήσει από τους 27 χώρες που μένουν πίσω να πληρώσουν την ύφη για κάποιον που θέλει να αποχωρήσει τώρα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ο τρόπος λοιπόν για να το κανονίσουμε αυτό είναι να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές λογιστικές και μετά αφού τις συμφωνήσουμε θα βγει το νούμερο στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Αλλά δεν είναι θέμα εκδίκησης ή τιμωρίας, δεν είναι σωστό και δίκαιο να το λέμε αυτό. στο ίδιο πλαίσιο δεν υπάρχει σταχυολόγηση, ε, το λεγόμενο cherry picking, δεν θα έχουμε ε, τέτοιες ε, σχέσεις, δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να βάλουμε στο πρώτη θέση τους πολίτες. Για το εμπόριο τώρα υπάρχουν κάποιες επίσημες κυρώσεις που δεν υφίστανται στην Βρετανική πλευρά ε, έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες διαπραγματεύσεις εμπορικές με τις ίδιες χώρες που έχουμε και εμείς διαπραγματεύσεις. Ε, έχουμε ήδη στο ψήφισμα δείξει και καταδείξει τι θα θέλουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν κάποια επίσημα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν δύσκολο να έχουμε, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο να διαπραγματεύεται με μια χώρα και ταυτόχρονα και εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να είναι ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είσαι ταυτόχρονα σε δύο τραπέζια. Έχουμε κάνει ε, ήδη μια πρόταση στο ψήφισμα γι' αυτό και θα έχει νόημα να μείνουμε πιστοί σε αυτό. Και το τελικό ερώτημα, το άρθρο 50. Κύριε Σέπφλιν. Ελπίζω ότι θα είναι η μοναδική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 50. Ποτέ ξανά στο μέλλον. Δεν θα υπάρξει πλέον το πρόβλημα, εάν δεν χρειαστεί να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και τόσο κακό αυτό το άρθρο, δεν είναι τόσο ακριβές, αλλά η έλλειψη ακρίβειας μας δίνει κάποια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει χρόνος ε, για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Φερχόφστατ και ελπίζω να σας βλέπουμε σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Σταγματικών Ίσης και πλίσμε Ίσως την έρξη δεν πραγματεύσω να ξαναλέω ο Φερχόφστατ. εκτός αν έχουμε διαφορετικά στοιχεία στην εντολή διαπραγμάτευσης, οπότε θα επανέλθω νωρίτερα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον καθηγητή Πογιάς Μαδούρο στις Βρυξέλλες. Επειδή ήταν εδώ, ε, εκμεταλλευόμαστε και εμείς την παρουσία του, παρέμεινε στις Βρυξέλλες και ήρθε ε, εδώ στην Επιτροπή μας, άρα δεν του πληρώνουμε και τα ε, διπορικά ή τη διενητέρηση του καθηγητού Μαδούρο. Πάντως σας ευχαριστούμε κύριε Μαδούρο που είστε εδώ και σας δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνει ε, η Επιτροπή τη δυνατότητα να σας μιλήσω για τις συνέπειες του Brexit, ιδίω ό,τι αφορά την ηθαγένεια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και επειδή ε, μου δώσετε τη δυνατότητα να ακούσω την προηγούμενη συζήτηση που ήταν πάρα πολύ συναρπαστική και μάλιστα ένιωσα ότι ε, ένιωσα τον περασμό να κάνω κάποια σχόλια, αλλά δεν ήταν ο λόγος ε, της παρουσίας μου αυτός εδώ. Αλλά σε ό,τι αφορά τη μηχανή του χρόνου και το άρθρο 50, εδώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Όταν εγκρίθηκε το άρθρο 50, κάθε ε, νομικός, ε, ιδίως ε, οι συνταγματολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 50 το θεωρούσαν ως όχι μια δυνατότητα αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά για να νιώθουν πιο άνετα να παραμένουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν ο στόχο του άρθρου, έτσι τον αντιλαμβανόμασταν και πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό, γιατί έτσι είχε παρουσιαστεί ιστορικά. Δηλαδή, ναι, μεν επισήμω ή τυπικά προβλέπεται η δυνατότητα αποχώρηση, ενισχύουμε δηλαδή τον εθελοντικό χαρακτήρα, τον προοριστικό χαρακτήρα τη συμμετοχή, άρα τα κράτη-μέλη ένιωθαν πιο άνετα να παραμείνουν. Αυτό ήταν ο στόχο. Αυτό το λέω για να ε, έχουμε όλοι στο μυαλό μας πόσο απρόβλεπτες επτός μπορεί να έχει ο νόμος. Ε, και αν δούμε το Brexit και περιμένουμε να δούμε και την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας, ε, τότε θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μέχρι τότε νομίζω ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ποια και αν είναι η έκβαση. Ε, η πρόγνωση γίνεται μόνο στο τέλος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, λέμε, στην Πορτογαλία. Το λέω και στο κύριο Περέα που είναι Πορτογάλος. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικέ και τα ζητήματα, πολύ σύντομα ε, θέλω να αναφέρω σε σχέση με την ε, προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ε, πολιτών και υπηκών και άλλων ευρωπαϊκών κρατών που ζουν, διαμένουν στην Ηνωμένο Βασίλειο, και να δούμε τι θα γίνει και τώρα και όταν φτάσει η στιγμή του Brexit ε, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Πρέπει να δούμε την ημερομηνία, τις προθεσμίες, ε, αλλά θέλουμε να δούμε τι γίνεται και με την προστασία των δικαιωμάτων ε, των Βρετανών υπηκών που θα παραμείνουν ή που διαμέσα και ιδίω τι θα γίνει μετά το Brexit. Τη συζήτηση αυτή θα ήθελα να την ε, συσχετίσω με την ευρύτερη συζήτηση ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την ε, έννοια, μάλλον για την έννοια της ηθαγένειας. Μια πρώτη στρατηγική είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ακόμα και αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Αυτή είναι μια πιο φυσική προσέγγιση, αν θέλετε, που βασίζεται στο να αποσυνδέσουμε τα δικαιώματα των ε, πολιτών, δηλαδή Βρετανών υπηκών που διαμένουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηκών τρίτων ε, χωρών, που διαμένουν, άλλων ευρωπαϊκών χωρών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα ακόμη και αν δεν έχουν τις αντίστοιχες ηθαγένειες μετά τον Brexit οι υπηκοευτοί ουσιαστικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια δέσμη ε, δικαιωμάτων, να την ορίσουμε αυτή τη δέσμη δικαιωμάτων που θα πρέπει να την χάνουν προστασία, ελεύθερη κυκλοφορία, δικαίωμα εγκατάσταση, κοινωνική προστασία κτλ. κτλ. Όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν είναι το ίδιο με την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και της ηθαγένειας. Αυτό δεν το εννοώ ε, ως συμβολική πολιτική και μόνο αναγνώριση που είναι και αυτό σημαντικό βέβαια, θα έχει και ευρύτερες επιπτώσεις. Γιατί, διότι ένα από αυτά που κάνει η ηθαγένεια είναι ότι δίνει ένα δυναμικό χαρακτήρα ε, σε αυτά τα δικαιώματα, σε αυτή τη δέσμη δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτήν. Ακόμη και τα δικαιώματα που υπήρχαν και είχαν δοθεί πριν την ύπαρξη της έννοιας της ηθαγένειας. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η έννοια, η ηθαγένεια δεν ε, έφερε μαζί της νέα δικαιώματα. Κάποια πολιτικά δικαιώματα ναι. Για τους μη οικονομικά ενέργους πολίτες προσέθεσε κάποια δικαιώματα, αλλά αυτό που έκανε κυρίως και κυρίως μέσω της νομολογίας του δικαστηρίου ήταν ότι επέκτηνε το πεδίο, ε, το εύρος των υφισταμένων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αν τα αποσυνδέσουμε λοιπόν τα δικαιώματα από την ηθαγένεια, θα χάσουμε. Έχουμε και τα πολιτικά δικαιώματα. Μπορώ να παραμείνω, αλλά πέραν αυτού υπάρχει αυτή η δυναμική που χάνεται. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι αναφέρουν αυτό το ενδεχόμενο, ιδίως για τους πολίτες ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως στους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν επί το παρόντος σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Βέβαια θα μπορούσε αυτό αφηρημένα να αφορά όλους τους πολίτες. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία πολιτών νομίζω που αναφέρει αυτή, αυτό το ενδεχόμενο το οποίο ποιο είναι να διατηρήσουν αυτοί οι πολίτες την Ευρωπαϊκή Θαγέννη. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει με τρεις ε, τρόπους. Η πρώτη πιθανότητα, δυνατότητα θα ήταν ε, ένα είδος συνδεδεμένης θαγένειας, associated citizenship. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί θαγένεια, δίνει η θαγένεια στου υπηκό του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμα και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια συνιστά ένα θεμελιώδη μετασχηματισμό της αρχής της ηθαγένειας ως είναι σήμερα, που είναι ένα παράγωγο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια απορρέει από την εθνική ε, ηθαγένεια, από την υπηκότητα, την εθνικότητα. Σημαντικό από πολιτική και συμβολική πλευρά και αυτό βέβαια δίνει και μια συνέχεια στη συζήτηση που γίνει και παλιότερα. Ότι θα μπορούσε η χορήγηση τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να είναι εξάρτητη από την ε, εθνικότητα, την εθνική υπηκότητα. Αλλά πρέπει να δούμε και ποιο είναι ο πολύ βασικό αντίκτυπο που θα έχει το ότι η κρατική, η εθνική υπηκότητα δίνει ε, το δικαίωμα για απόκτηση ευρωπαϊκής ηθαγένειας είναι κάτι σημαντικό. Το αν όμως υπάρχει, αν θέλετε, φορητότητα αυτής της ηθαγένειας και πέραν των συνόρων του κράτους, ενισχύει ταυτόχρονα και τις σχέσεις με, με το κράτος, γιατί είμαστε ε, Ευρωπαίοι υπήκοοι, γιατί έχουμε ε, την υπηκότητα μιας χώρας μέλους της Ένωσης. Άρα έχει και θετικά και αρνητικά το να ανοίξουμε το παράθυρο ε, ή την πόρτα <laughs> σε αυτή την δυνατότητα. Μια άλλη επιλογή ενδεχόμενη είναι να γίνει μια συμφωνία σε πρώτο Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιβάλλει στα κράτη-μέλη να δίνουν στου ε, πολίτε από την Βρετανία που διαμένουν στο εδαφό του σε την ε, υπηκότητα τη χώρα στην οποία διαμένουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα καθορίσει του όρου χορήγηση ηθαγένεια υπηκότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι εφικτό και από πολιτική πλευρά. Και όπω και με την προηγούμενη εναλλακτική, για τι δύο αυτές αναλλακτικές απαιτείται αλλαγή τη συνθήκη, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση επί το παρόντο. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα που μπαίνει σε αυτή την αποσύνθεση των δικαιωμάτων που δεν σχετίζονται με την ηθαγένεια. Δηλαδή, οι Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν σε άλλα κράτη-μέλη θα έχουν ε, μια δέσμη δικαιωμάτων που σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαίοι υπήκοοι. Μία από τις διαφορές σε ό,τι αφορά το καθεστώς ενός υπηκόου ε, ευρωπαϊκής χώρας που θα συνεχίσει να διαμένει στο Ηνωμένο και τις σχέσεις, ή μάλλον τις, ε, του καθεστώτος ενός Βρετανού υπηκόου που ζει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχουν βρετανικό το δικαίωμα διαμονής και να έχουν κάποια παράνομα δικαιώματα, αλλά χάνουν μια σημαντική διάσταση της κινητικότητας δηλαδή. Δεν μπορούν οι Βρετανοί να μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Βέβαια με το άρθρο 79 μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, γιατί έχει την νομική βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίσει με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματα των επικών τρίτων χωρών που, κατοικούν, που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Όμως, πάντα γυρίζοντα πίσω στην ε, πιθανότητα, να, στη δυνατότητα να αποσυνδέσουμε τα δικαιώματα από τα ηθαγένεια. Και υπάρχει και μία άλλη ε, επιλογή, μια άλλη εναλλακτική που δεν είναι καθόλου πιθανή κατά την απόψή μου και είναι αμφίβολη και απονομική νομική, αμφίβολη πλευράς και θα είναι πρόκληση και για το δικαστήριο. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ε, στην, υπόθεση Ρότμαν η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου που ήταν ε, ο γενικός ε, εισηγητής του δικαστηρίου στην προκειμένη περίπτωση τότε για πρώτη φορά το δικαστήριο, συγκεκριμένη απόφαση του λέει ότι ακόμη και αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει σε ένα κράτο μέλο του όρου για την απόκτηση, την απώλεια μια εθνική εθνικής υπηκότητα, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει ή να ελέγξει του όρου από του οποίου τα κράτη-μέλη αποσύρουν την ηθαγένεια ενό ε, υπηκότου. Και λέει το δικαστήριο ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ορίσουν την απώλεια ε, της ηθαγένειας κατά δυσανάλογο τρόπο. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όταν κάποιοι προσβάλλουν την απώλεια ηθαγένειας λόγω Brexit, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ομολογία ερώτημα και να πούν ότι θα είναι δυσανάλογο κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι πιθανό βέβαια να επιτύχει κάτι τέτοιο, διότι εάν το δικαστήριο ε, το υποστηρίξει αυτό, τότε στερεί οδήποτε νοήματος ε, το άρθρο 50. Αφού αν κάποιος αποχωρεί χάνει και την ηθαγένεια. Άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε και να συμφιλιώσουμε αυτούς τους δύο στόχους. Βέβαια υπάρχει μια οπτική γωνία για αυτή τη νομική πρόκληση ε, που θα μπορούσε να επιτύχει με αυτόν τον τρόπο αυτή η πρόκληση. Νομίζω ότι ετέθη πριν το δημοψήφισμα το ζήτημα, ξέρω γνωρίζω, και πρέπει να πω ότι τότε εγώ νόμιζα, ή τέλο πάντων είχα καταλάβει, γιατί από πολιτική πλευρά δεν προχώρησαν με αυτό. Ίσως ε, και γι' αυτό δεν απευθύνθηκαν ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα Βρετανικά δικαστήρια για το θέμα αυτό. Από νομικές πλευράς όμως υπήρχε ένα βάσιμο επιχείρημα, το οποίο είναι το εξή. Αν οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Πολλοί δεν είχαν δικαίωμα ψήφου στο δημοψήφισμα. Νομίζω θα έχουν ένα πιο ισχυρό επιχείρημα για να επικαλεστούν τον τρόπο με τον οποίο θα απολέσουν την ηφαγένεια, την ευρωπαϊκή υφαγένεια. Ουσιαστικά είναι υποχρεωμένοι, τους επιβάλλεται να απεμπολίσουν την ηθαγένεια, χωρίς όμως να είχαν μπορέσει να εκφράσουν προηγουμένως την άποψή τους. Δεν είχαν φωνή, δεν είχαν ψήφο. Αυτοί μπορούν, πιστεύω, να προσβάλλουν την απόφαση. Δεν σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει. Όμως, ακόμα και απόφαση ένα κράτος μέλους να αποχωρήσει πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κάποιες θεμελιώδεις αρχές, μία από τι οποίε είναι για παράδειγμα το δικαίωμα συμμετοχή όλων των υπηκών αυτού του κράτου μέλους να μην στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής ε, στη διαδικασία λήψης απόφαση επειδή διαμένουν σε ένα κράτος μέλος. Να είναι αυτός ο λόγος. Είναι πολύ σημαντική η πτυχή αυτή. οικονομικής πλευράς νομίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Από πολιτικής πλευράς αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι είναι άκρο απίθανο ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δεχθεί ε, να την, την επιχειρηματολογία αυτή, αλλά είναι, είναι μια ε, βάσιμη επιχειρηματολογία. Μια άλλη εναλλακτική είναι κάποιοι Βρετανοί πήκοοι να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή Θαγή και άλλοι όχι. Αυτό θα είναι ένα, είναι ένα πρόκλησης. Τίποτα δεν εμποδίζει ένα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνει και ένα άλλο τμήμα να αποχωρήσει και έχουμε ένα προηγούμενο που λέγεται Γρυλανδία. Δηλαδή έχουμε την, υποθε... την περίπτωση ενός κράτου μέλου όπου ένα τμήμα τη επικράτειά του εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα άλλο παρέμεινε. Επομένως, ε, ε, επί της αρχής δεν αποτρέπει τίποτα, ε, παραδείγματο χάρη τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία, να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη επικράτεια του Νομίου Βασίλειου να μην ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό θα είναι πάρα πολύ πολύ να δει στην πράξη, διότι θα απαιτεί εσωτερικά σύνορα μέσα σε μια χώρα, μέσα στην ίδια χώρα σε σχέση παραδείγματο χάρη με την ε, Ιρλανδία και τη Βόρεια Αλλά από πολιτικής πλευρά είναι άκρο προβληματικό και υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες καθιστούν κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο. Ένα κίνδυνο θα ήταν οικονομικό για τον Ηνωμένο Βασίλειο, διότι για τη Σκωτία και τη Βορειολλανδία θα είναι πάρα πολύ θετικό βέβαια γιατί θα προσελκύσουν πάρα πολλέ επενδύσει και πολλέ επιχειρήσει που θα μετεγκατασταθούν στι περιοχέ αυτέ γιατί μπορούν να αποφεληθούν από τι αγορέ του. Βέβαια, για το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δραματική γιατί θα υπάρξει οικονομική κινητικότητα μετατόπιση προ αυτέ τι δύο περιοχέ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυσκολία θα είναι ότι αν αυτό γίνει χωρίς επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως κράτους, εφόσον μέρος του κράτους θα παραμείνει, μέρος σε θα παραμείνει, όπως ε, συνέβη με Δανία, Γρυλανδία, αυτό τι θα σημαίνει. Η εκπροσώπηση του τμήματος αυτού της επικράτησης θα γίνεται από τη Βρετανική κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις Σκοτίας και Βορειολανδία. αν δεν αποχωρήσουν και ξαναμπούν ως Σκοτία Warriors, δηλαδή οπότε και έχουμε απόσχηση, αν δεν γίνει αυτό τότε θα πρέπει ε, η κεντρική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου να εξακολουθεί να έχει την ε, ευθύνη. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα να φύγει η χώρα ως Ηνωμένο Βασίλειο και να μπουν μετά ως τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι μια εναλλακτική. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων υπηκών ε, στη... στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν σημαντικά θέματα. Ποια είναι η προθεσμία πρώτα απ' όλα. Η κατάληκτη ημερομηνία. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μένουν στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο, ποια είναι η προθεσμία που πρέπει να πάρουμε όσον αναφορά. η ημερομηνία του δημοψηφίσματο, η ημερομηνία ολοκλήρωσε της συμφωνίας, η νέα συμφωνία Brexit, ε, πότε θα υπογραφεί ή πότε θα αρχίσει να ισχύει, πότε θα τεθεί σε ισχύ, αν δεν συμπέσουν αυτά τα δύο. Κατά την άποψή μου. Πριν από την ημερομηνία του ίδιου του Brexit, αν βάλουμε την ημερομηνία, ήδη περιορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είναι ακόμα μέλος ε, της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή αν πούμε ότι θα προστατεύσουν τα δικαιώματα μόνο αυτών οι οποίοι θα ζουν, μέχρι, ζούσαν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τη μέρα του δημοψηφίσματο ή μέχρι τη μέρα που κατατέθηκε ε, το αίτημα δυνάμει του άρθρου 50. Είναι σαν να λέμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφούται ήδη από τότε προς κάποιες από τις υποχρεώσεις που υπέχει λόγω της συμμετοχής στην Ένωση. Άρα εγώ νομίζω ότι η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι η η ημερομηνία της πραγματικής ε, αποχώρησης και το πολύ ημερομηνία υπογραφής συμφωνία. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα μάλλον ε, ροής ε, μαζικών ροών ανθρώπων για να αποφύλλονται των δικαιωμάτων που δεν είναι μεγάλη βέβαια πιθανότητα. Υπάρχει όμως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο μηχανισμός που θα μπορούσε να το αποτρέψει. Έχει πει το δικαστήριο σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ότι αν είναι τεχνητή αμυγός αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία δεν, είναι, δεν αναγνωρίζεται γιατί θεωρείται απάτη ουσιαστικά. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το επιχείρημα από το δικαστήριο. Και είναι και το πιο σωστό. Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Η νομική προστασία και η ερμηνεία των δικαιωμάτων αυτών μετά την αποχώρηση του Βασιλείου. Εδώ ευθυγραμμίζομαι σε μεγάλο βαθμό με το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών που είχατε δυνατότητα να μελετήσω. Στον γραφό αυτό της Κομισιόν προτείνεται ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που ισχύει στον ΕΟΧ, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να δεσμεύεται από την ε, προηγούμενη νομολογία και απαιτείται να λαμβάνει υπόψη του στο μέλλον και την νομολογία του ε, δικαστηρίου για αυτά τα δικαιώματα τα οποία θα διατηρήσουν να έχουν αυτοί που θα συνεχίσουν να παραμένουν, να διαμένουν στον Ευρωπαϊκό και αντιστρόφως για τους Βρετανούς πικούς που θα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη έχουμε και τα θέματα της ΕΖΕΣ όπου δεν θεωρεί ε, το δικαστήριο της ΕΖΕΣ ότι θα πρέπει να δεσμεύονται οι χώρες για το μελλοντική νομολογία. Θα πρέπει να την εφαρμοσει Το θέμα είναι δικαστήριο, ποιο δικαστήριο θα εφαρμόσει αυτή την ε, νομοθεσία. Γιατί όχι τα βρετανικά δικαστήρια. Δεν θα είχα ιδιαίτερε επιφυλάξει γιατί το βρετανικό νομικό σύστημα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης έχει δείξει ότι είναι πιστό στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και πολύ περισσότερα από άλλες δικαιοδοσίες μάλιστα. Άρα εγώ εμπιστεύομαι τα βρετανικά δικαστήρια για να εφαρμόζουν και να ε, επιβάλλουν το σεβασμό αυτών των ε, δικαιωμάτων. Ε, στην ΕΖΕΣ η εφαρμόζεται από τον ΕΟΧΟ. Εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα. Θα εφάρμοζα ένα αντίστοιχο μηχανισμό και δεν θα δημιουργούσα ένα νέο δικαστήριο για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Μια ερώτηση πριν να κλείσω, μάλλον ένα θέμα πριν να κλείσω. Το ένα σχετίζεται με αυτήν την ευρύτερη έννοια της ε, ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαίου πολίτη. Πιστεύω πως ε, η απώλεια της ε, δημοφιλίες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το Brexit ε, οφείλεται στο ότι ε, υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικές απόψεις των πολιτών και οι πολίτες ακολουθούν θέσεις ανάλογα με το αν είναι κινούμενοι ή μη κινούμενοι οι πολίτες. Υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι είναι κινούμενοι και, και ότι είναι κομμάτι ενός ανοιχτού κόσμου που χρησιμοποιούν την κινητικότητά τους και ακόμα και όταν πραγματικά δεν κινούνται η κατανόηση του κόσμου ε, που έχουν ε, καθορίζεται από αυτό το μοντέλο και έχουμε μια άλλη ομάδα πολιτών που δεν είναι κινούμενοι και που έχουν την αντίθετη εικόνα του κόσμου ως προς αυτό. Είναι πιο στατική. Ε, κάτι που μπορούμε να μάθουμε λοιπόν είναι ότι ένα από τα προβλήματα ή ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη είναι ότι θεωρείται αυτό θετικό μόνο από αυτούς που θέλουν να κινηθούν, ενώ οι στατικοί θεωρούν ότι είναι ξένοι προς την έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και των ε, ωφελών της, και των της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε <coughs> τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής ηθαγένειας να καταστούν σαφέστερα σε αυτό το, σε αυτό τους τους πολίτες τους πιο στατικούς. Κάτι ακόμα που μπορεί εξ αρχή να φαίνεται παραδοξικό. Ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένεια είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται ε, στιάζεται στους λευκούς. Δεν έχεις πολίτες παρά μόνο όταν, ε, συγγνώμη, ε, στιάζεται στα δικαιώματα και όχι στα, υποχρεώσει. Και οι πολίτες δημιουργούνται μόνο εφόσον κατανοήσουν ότι έχουν μεν δικαιώματα, αλλά ότι έχουν και υποχρεώσεις, καθήκοντα. Και αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από πέντε χρόνια το τόνισε αυτό σε μια έκθεση προς το, εδώ το Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει και συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Είναι μια παλιά μου μανία ε, ότι ε, αυτό το θέμα που θα μετατρέψει όλα τα ζητήματα και θα αλλάξει όλες τις οπτικές για όλα τα θέματα είναι ε, το θέμα των ιδίων πόρων. Αυτό είναι ένα δηλητηριώδες θέμα και ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί η Ένωση είναι λάθος γιατί δεν καθιστά σαφές στους πολίτες ότι οι ίδιοι φέρουν το φορτίο, δεν καθίσταται σαφές ποια είναι τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μετατρέπει οποιαδήποτε συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι που στην ουσία καταλήγει σε ισοπαλία ή μηδενικό αποτέλεσμα. Πάντως, θα έχουμε μόνο να κερδίσουμε αν σχεδιάζοντας τους ίδιους πόρους και συνδέοντας αυτούς τους ίδιους πόρους με μια κατανόηση από πλευρά των πολιτών ότι μοιράζονται το φορτίο και πώς το μοιράζονται και επίσης συνδέοντας πάλι ε, ε, το θέμα των ιδίων πόρων με τα ωφέλη ή με τα θέματα φορολογίας, τα κομμάτια της φορολογίας που οι, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν πλέον να, να επιβάλλουν τα ίδια. Και έτσι θα έχουμε και τους πολίτες που θα λέμε και θα τους πούμε ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι που τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να το κάνουν. Επαναφέρει τη δικαιοσύνη στη φορολογία όταν τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό κατά τη γνώμη μου αυτό. Τέλος. Που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον Brexit, αλλά συνδέεται και με τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ίσως να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πόσο το Brexit θα πρέπει να συνδεθεί με τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι μια επανάληψη της συζήτησης που έγινε πριν από το δημοψήφισμα. Εάν θυμάστε, όταν συζητήθηκε το ειδικό καθεστώς για το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να αποφευθεί μάλιστα τότε το Brexit, ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Ας το κλείσουμε όσο γίνεται το θέμα, να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική κατάσταση για να μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Δεν δούλεψε. Απέτυχε. Και η γνώμη μου είναι ότι είναι ίσως καλύτερα να το συνδέσουμε με την ευρύτερη συνταγματική συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τρεις λόγους. καταρχάς γιατί ό,τι και αν αποφασίσουμε για το Brexit θα χρειαστεί ομοφωνία και επικύρωση από όλα τα κρατημέλη. Μάλλον. Ενώ το άρθρο 50 όχι. Είναι ειδική πλειοψηφία αλλά αν δεν υπάρξει πραγματικά, πραγματικά σκληρό hard Brexit και αυτό θα ήταν πολύ κακό πιστεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δραματικό για το Ηνωμένο Βασίλειο, πάντως εάν δεν συμβεί αυτό, τότε οποιαδήποτε συμφωνία για το Brexit υπό το άρθρο 50 θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση μιας νέας συμφωνίας, σύναψη μάλλον μιας νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο που πιθανότατα θα απαιτήσει την ομοφωνία και την επικύρωση από τα κρατημέλη. Εάν λοιπόν πρέπει ούτε κανείς να κάνει αυτή τη διαδικασία, να περάσει από αυτή τη διαδικασία, θα, πρέπει να το κάνει μαζί ως ένα τμήμα των, ε, ε του ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων. Ε, και τέλος, δεν αποκλείουμε τη δυνατότητα να βρούμε μια τελική λύση όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει και θα μείνει ταυτόχρονα. Εάν έχουμε δηλαδή μια, ευρύτερα μια Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικούς κύκλους ολοκλήρωσης, κανέ, τίποτα δεν εμποδίζει αυτή η εναλλακτική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί έναν από τους κύκλους ολοκλήρωσης και έτσι θα υπάρχει δυνατότητα το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο να βγει και να ταυτόχρονα μείνει. Αλλά με πιο αδύναμη μορφή ένταξη. Αυτό σημαίνει βέβαια την αποδυνάμωση συνταγματικών, ε, σημαίνει μάλλον κάποιες συνταγματικές τροπολογίες και νομίζω ότι το άλλο δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν το συζητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης δημοκρατικό έλμα όταν δεν μπορείς συνταγματικά να τροποποιήσεις τον εαυτό σου. Γιατί οι νέες γενιές οφείλουν να δεσμεύονται από αυτά που αποφασίστηκαν στο παρελθόν. Κατανοώ τις δυσκολίες και γιατί κανείς δεν θέλει να ανοίγει νέα διαδικασία με τροποποίηση των συνθηκών και εγώ ίδιος το υποστήριζα αυτό χρόνια και χρόνια όταν καλύτερο να μην αρχίσουμε μεγάλη συνταγματική συζήτηση και να προσπαθήσουμε ε, συνταγματικά να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί όμω να μεταρρυθμίσουμε τη συνθήκη, δηλαδή να βρούμε μια ερμηνεία από το δικαστήριο, αλλά πιστεύω πω είναι και πλέον η ώρα να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα. Πριν από κάποια χρόνια, μαζί με έναν συνάδελφο από το Yale, προτείναμε κάτι που ονομάσαμε ε, Νότια πρόταση. Και την επαναλαμβάνω, γιατί την είπαμε έτσι, γιατί στην Νότια Αφρική είχαν ένα παρόμοιο πρόβλημα με το τέλος του Απαρτχάιντα. Ήθελαν ένα σύνταγμα που θα, που θα αντικατόπτριζε τα συμφέροντα και όλων το... της πλειοψηφίας του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα θέλανε κάτι που θα μπορούσε να γίνει δεκτό από όλες τις διαφορές ε, κοινότητες, τις αρχές της ε, μεταρρύθμισης. Οπότε, συμφώνησαν καταρχάς για έναν χάρτη βασικών αρχών, στον οποίο θα μπορούσε να βάλει βέτο οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες και έπειτα το Σύνταγμα έπρεπε να ε, είναι σύμμορφο προς αυτό το χάρτη. Και η ε, ε, συμμόρφωση προς αυτές τις βασικές αρχές ελεγχόταν από το νέο συνταγματικό δικαστήριο. Να έχουμε δηλαδή και εδώ μια διακυβερνητική διάσκεψη που θα αποφασίσει μόνο για ένα, μια, ένα γενικό σύνολο κανόνων και ε, επίσης ε, μετά να συνταχθεί ένα λεπτομερές έγγραφο έτσι ώστε ταυτόχρονα να πρέπει να κυρωθεί το έγγραφο των βασικών αρχών και το λεπτομερές έγγραφο και η συμμόρφωσή του με τις βασικές αρχές θα ελεγχθεί από ένα ad hoc δικαστικό σώμα που θα αποτελείται από τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστήριων των διαφόρων κρατών μελών. Αυτό ήταν μάλλον ένα τρόπο για να μπορέσουμε να λύσουμε τα χέρια, το γόρδιο δεσμό. Δεν ήταν εύκολο, το καταλαβαίνω, αλλά πάντως θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε όσον αφορά την τροποποίηση των συνθήκων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέσατε των δάκτυλο επί των τύπων των ύλων σε πολλά ζητήματα. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν οι ερωτήσει. Η Βάρμπαρα έχει σηκώσει το χέρι και μετά ο Σα Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα διήγηση σε σχέση με τα δικαιώματα. Αυτό που θέλω... Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι αυτό που είπατε για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, δηλαδή ως ένα δικαίωμα για τον κινούμενο ε, ε, πολίτη και όχι για τον στάσιμο. Συμφωνώ απόλυτα για το ζήτημα το κρίσιμο των ίδιων πόρων, που εάν ε, αυξηθούν θα έδιναν την εντύπωση μεγαλύτερη συμμετρίας και αλληλεγγύης στην Ένωση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως ε, είναι από την άποψη που τι θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή τις διάφορες μορφές ηθαγένειας ή δικαιωμάτων συνδεόμενων με την ηθαγένεια. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση για τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πιστεύετε πως είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το σύνθημα που διαρκώς επαναλαμβάνεται από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την προδιαπραγματευτική διάδικα... Ε, περίοδο, ότι δηλαδή ε, δεν θα είναι καλύτερα εκτός της Ένωσης η Εγγλέζοι. Είναι κάτι που το ακούμε και ξανά μανά και το μας, αρχίζουμε να το συνηθίζουμε. Αλλά είναι ένα είδο μεγάλη απειλή. Δεύτερον, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι καλύτερα έξω από ότι μέσα στην Ένωση. Και δεν έχουμε, δεν είμαστε βέβαιοι 100%. Ευχαριστώ. Thank you, Mercedes. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Mercedes Μπρέσο. Καταρχάς, ναι, ναι, αυτό που ε, λέει η Μπάρμπαρα δεν είναι πολύ είναι αλήθεια, γιατί δεν τους λέμε αυτό. Λέμε ότι... Ε, ε, μπορεί κανείς να μείνει μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Εκεί είναι πρόβλημα αυτού που βγαίνει. λοιπόν, εγώ μπορώ να κάνω είναι να ρωτήσω σε εσά, Πρόεδρε, αν κάποια άλλη στιγμή, γιατί εδώ βεβαίω μιλάμε για το Brexit, αλλά μήπω θα μπορούσαμε για την εμβάθυνση που θα κάνουμε για αυτό το θέμα των δικαιωμάτων των ε, πολιτών, που το κάνουμε και για την κοινωνική Ευρώπη, μήπω θα έπρεπε να σκεφτούμε ε, αυτό το θέμα για περισσότερο χρόνο, δηλαδή να έχουμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε, γιατί Π.χ. στη συζήτηση των ημερών για το θέμα των αποσπασμένων ε, εργαζόμενων. Μήπως αυτό θα μπορούσε να είναι κατάχρηση του δικαιώματος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας για ανθρώπους που κινούμενους, μετακινούμενους σε σύγκριση με τους στάσιμους. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα μπορούσαν αυτά να μας χρησιμεύσουν και για το Brexit, γιατί στο μέλλον το πλαίσιο των σχέσεων και για τους πολίτες θα πρέπει να είναι καθορισμένο. Θα πρέπει δηλαδή να εμβαθύνουμε πολύ καλά στο θέμα αυτό της κινητής ή ακίνητης ηθαγένειας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά κατά τη γνώμη μου. Τελευταίο μου ερώτημα για το θέμα της Ιρλανδίας και της Σκοτίας. Αν κατάλαβα καλά, Εσεί θεωρείτε πω είναι δυνατόν να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία αν το αποφασίσουν μέσω δημοψηφίσματος π.χ. παραδείγματο χάρη χωρί να υπάρχει επίσημη έξοδο και εκ νέου είσοδο, Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να μπουν αλλά να εκπροσωπούνται από τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα και αν δεν ήταν κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή η υπόθεση ότι μπορεί απλά χωρίζοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνουν στην Ένωση θεωρείτε πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Είναι πιο ξεκάθαρο να βγουν και να ξαναμπούν με την προπόθεση ότι θα είναι γρήγορη η διαδικασία. Γιατί ήδη έχουν ε, σε εφαρμογή το κοινωνικό κεκτημένο, ε, αν και νομικό νομικός ω νέο κράτο θα έπρεπε να δεχτούν όλη το νέο, την νέα αυτή νομοθεσία το κοινοτικό κεκτημένο. Εν πάση περιπτώσει αυτό ε, το ρώτησαν οι εκπρόσωποι της Σκωτίας, που θέλουν να κατανοήσουν ποια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσουν αν αποφασίσουν να αποκοπούν από το Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο να μείνουν στην Ένωση. Και μια ερώτηση όσον αφορά την Ιρλανδία. Μάλλον πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση εκεί. Τι, ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ ευχαριστώντας ε, τον κύριο Μαντούρο για την παρουσίαση. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Βέβαια όλοι είμαστε σε αυτή την ε, φάση που προσπαθούμε να ελέγξουμε τις ε, ζημίες. Όμως ε, το Brexit θα έχει επιπτώσεις και ως προς τα δικαιώματα των πολιτών και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια κατανοείται ως μια πολυεπίπεδη ηθαγένεια όπως την έχουμε στις συνθήκες. Βέβαια, υπάρχει μόνο για τους πολίτες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι εναλλακτικέ είναι μάλλον οράματα, παρεσθήσεις. Ε, οποιαδήποτε περίπτωση ε, πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή έκβασή της. Τώρα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δικαιώματα της ε, διαμονής και το τι μπορούμε να κάνουμε για να τα προστατεύσουμε στο μέλλον. Τώρα, ένα από τα πράγματα, ε, μία από τις συζητήσεις αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ζητά πολλά χαρτιά από τους μετανάστες για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα παραμονής, 80 σελίδες ας πούμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα υφιστάμενα δικαιώματα διαμονής που έχουν οι πολίτες που ήδη ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ κλείνει η συζήτηση ε, και γι' αυτό δίνω το λόγο στον κύριο ε, Μαντούρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω και σε αυτή την τελευταία ερώτηση σίγουρα. Το ευρωπαϊκό δίκαιο ως έχει τώρα και οι διαδικασίες είναι δηλωτικές και όχι ε, διαδικασίες που δημιουργούν τα δικαιώματα. Άρα οι διαδικασίες πρέπει να είναι όσο πιο απλές γίνεται. Αυτά τα ε, δικαιώματα ως ισχύουν αυτή τη στιγμή ε, οποιαδήποτε γραφειοκρατία που ακούμε όπως ας πούμε το να πρέπει κανείς να συμπληρώσει 80 σελίδες όλα αυτά θα, μπορούν, θα αποτελούν παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Αν έχουμε λοιπόν απλώς το δικαίωμα παραμονή στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να παραμείνει και να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον τρόπο που έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οτιδήποτε άλλο θα είναι παράνομο. Αν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδό του αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο, θα έχουν δικαίωμα προσφύγης στο δικαστήριο. Ε, η απάντησή μου είναι ότι ε, εμπιστεύομαι τα αγγλικά δικαστήρια, τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι θα εφαρμόσουν αυτά που έχει ήδη αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε παρόμοιες υποθέσεις. Θα υφίσταται δηλαδή με την ερμηνεία και τις εγγύησεις που συνδέονται με αυτό το δικαίωμα πριν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ε, οι αρχές αυτές δεν δημιουργούν το δικαίωμα, είναι δηλωτικές. Και τώρα η νομική εφαρμοσιμότητα και νομική προστασία είναι ένα άλλο θέμα Κατά την άποψή μου θα αρκούσε να πω ότι τα Βρετανικά δικαστήρια θα το κάνουν αυτό διότι δεσμεύονται από τις ε, προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους ε, στο μέλλον. Τώρα για τους κινητούς και μη κινητούς πολίτες, κινούμενους και μη κινούμενους πολίτες. Αν δούμε όλα τα όσα έχουν συμβεί, και πώς εξελίχθηκε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, ήταν ε, μια διαδικασία κρίσιμη όλη αυτή. Ε, είχαμε τους μη οικονομικά ενεργούς πολίτες και το δικαίωμα κινητικότητας αυτών. Δεν το συζητήσαμε πολύ, αλλά όταν μιλήσαμε για τη μελλοντική συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και όταν ακούμε τη σημασία διατήρησης της ακαιρεότητας της εσωτερικής αγοράς και της ελεύθερης κίνησης, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα κατά την άποψή μου είναι μιλάμε μόνο για οικονομικά ενεργούς πολίτες ή και για τα δικαιώματα αυτών που δεν είναι ενεργοί οικονομικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε. Και αυτό που είναι ακόμα πιο κρίσιμη σημασία είναι ότι τελικά θα πρέπει να έχουμε εργαλεία τα οποία θα μας δείξουν τι σημαίνει ευρωπαϊκή ηθαγένεια ακόμα και για αυτούς που δεν κινούνται. Επίσης, η σχέση με τους ίδιους πόρους είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή υποθετικά απλώς το συζητάμε Ας πούμε, ε, το Ταμείο Ανεργίας ε, για την απορρόφηση ασύμετρων, κραδασμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία στην ε, περιοχή του ευρώ, στον χώρο του ευρώ, όλα αυτά είναι μια προστασία για τους πολίτες. Για τις διαπραγματεύσεις να πω ότι θεωρώ πως πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκολία των ίδιων των διαπραγματεύσεων. Πρέπει αυτό να το περιορίσουμε με ένα φυσικό τρόπο. Και εγώ δεν έχω εμπειρία ε, με διαζύγιο, ούτε και με γάμο δεν έχω. Προσπαθώ να αποφύγω οτιδήποτε ενέχει περίπλοκες συναλλαγές και κόστη. Είναι φυσικό όμως η ίδια η διαδικασία να κάνει την διαπραγμάτευση ακόμα πιο δύσκολη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι σημαντικό να το αποφύγουμε και αυτό. Κατά την άποψή μου, ο τρόπος που πρέπει να το κάνουμε είναι να πούμε Εντάξει, είναι προβληματικό να πούμε στους ε, Βρετανούς εκ των προτέρων ότι θα είμαστε πιο μαλακοί από, ε, θα, θα είστε πιο μαλακοί από ό,τι πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους πούμε τίποτα, ας το αποφασίσουν αυτοί, γιατί αν το κάνουμε θα το αντιληφθούν διαφορετικά. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη κίνηση. Αυτό είναι πλήρως αποδεκτό. Τώρα το να προσθέτουμε επίθετα και προσδιορισμούς σε όλα αυτά ε, δεν βοηθά σε καμία περίπτωση. Για τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκοτία. Δεν αποκλείω την πιθανότητα να αποφασίσουν η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία να αναξαρτητοποιηθούν αν γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα ανεξάρτητα μέλη. Αυτό δεν είναι νομικά αδύνατο, πολιτικά θα πρέπει να το δούμε. Αλλά τι λέω ότι υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική που έπεσε στο τραπέζι εάν μείνουν η Βόρειος Ιρλανδία και η Σκοτία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να παραμείνουν και ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο τρόποι νομικά να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, να πούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν φεύγει, μόνο κομμάτι της επικράτειάς του, όπως έγινε με τη Γρυλανδία και τη Δανία. Να υπάρχει λοιπόν μια διαδοχή και Αυτό ε, είναι το, ένα ζήτημα. Τι κάνουμε όταν έχουμε μια συμφωνία με ένα κράτος μέλος που φεύγει αλλά μέρος της επικράτειάς του παραμένει όπως έγινε με τη Δανία και τη Γρινλανδία. Αν γίνει έτσι, η επιπλέον δυσκολία που εγείρεται είναι ε, ότι αυτός που μένει είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ως Ηνωμένο Βασίλειο και η αντιπροσωπεία του ε, στο Συμβούλιο και τα λοιπά ή εσωτερικά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναδιοργανωθεί και να πει ότι εμείς αναθέτουμε την εκπροσώπησή μας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, στη κυβέρνηση της Σκοτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Η δυσκολία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το σημείο είναι ότι τελικά αν το κάνουμε έτσι θα παραμείνει ως δούριος ύπος το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα το αντιληφθούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Να φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο και μέρος του να μένει με νέα συμφωνία. Να έχουμε δηλαδή τη Σκοτία και την Ιρλανδία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να είναι και μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό να νομικά είναι διαφορετική εναλλακτική. Ευχαριστώ. Very much. It was extremely useful. Uh, thank you. Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε κύριε καθηγητά. Ελπίζω πριν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία να έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναέχουμε εδώ. Oh, I'm sorry, I didn't notice. Yeah. Δεν σας ε, ε, πρόσεξα κύριε Φόξ. Ε, παρακαλώ το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο μα μας ε, κάπως τα μπέρδεψε στα τελευταία σχόλια που έκανε, γιατί μιλήθηκε, μίλησε συγγνώμη, για ανεξαρτητοποίηση Σκοτίας Βορειοϊρλανδία. Προς ενημέρωσή σας. Κανένας δεν λέει η ε, να γίνει ανεξάρτητη. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Δημοκρατίας Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου ότι οι Βορειοϊρλανδοί θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο θα παραμείνουν ε, τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου ή θα προσχωρήσουν στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Η συνέλευση της ε, Βόρειας Ιρλανδίας ε, θα οργανώσει τη σχετική διαδικασία. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί ήταν ανακριβές αυτό που είπατε. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον Πασκάλ Ντυρά. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Λοιπόν, κανό και γενικέ αρχέ για σχετικά με του τρόπου ελέγχου από τα κράτη-μέλη τη άσκηση των τελικών αναμετρών από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βιάζομαι λίγο, γιατί παράλληλα υπάρχει μια συνδρέση και ε, στην οποία πρέπει να πάω και ήθελα να προλάβω η ανταλλαγή απόψεων πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα και αφορά το θέμα της επιτροπολογίας και συγκεκριμένα για την εκτελεστότητα ε, δεσμευτικών πράξεων. Έχουμε μια πρόταση της Κομισιόν για να προσπαθήσουμε να βγούμε από τη δυσχερή θέση που αντιμετωπίζει η Κομισιόν, που είναι και πολιτική και αφορά και τις σχέσεις ε, με τρίτους, με συμβαλωμένους, ε, συγκεκριμένα. Σε μια διαδικασία εξέτασης, όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία δεν μπορεί η Κομισιόν ούτε να εγκρίνει ούτε να απορρίψει την εν λόγω πράξη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μια απόφαση. ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, κάτι που δυσκολεύει τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να υποκαταστήσει τα κράτη. Υπάρχουν προτάσεις λοιπόν που γίνονται από την Κομισιόν. Πρώτη είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε απλή διαδικασία και μετά έφεση εντό αγωγικών και έπειτα θα μπορούσε να προσθεθεί και μια δεύτερη στην έφεση. Αν ε, πρωτοβαθμίως επιβεβαιωθεί ε, αυτό που έχει αποφασιστεί, ε, το να προσθέσουμε ένα τρίτο επίπεδο ε, γίνεται πιο δυσκίνητη όλη η διαδικασία γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι στο τρίτο βάθμιο επίπεδο θα ακυρωθεί απόφαση των δύο πρώτων βαθμών, βαθμίδων. Μια άλλη πρόταση της Κομισιόν μου φαίνεται μάλιστα ότι είναι και πιο επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, είναι να μειωθεί απαρτία για την έφηση. Δηλαδή να έχουμε απλή πλειοψηφία και να μην λαμβάνονται πλέον οι αποχές υπόψη, να μην τις μετράμε. Άρα μειώνουμε την απαρτία και από ένα σύστημα ειδικής πλειοψηφίας περνάμε σε ένα σύστημα απλής πλειοψηφίας. Άρα τα κράτη-μέλη ουσιαστικά τα βολεύει να μην αποφανθούν, γιατί μετά μπορούν να απαλλαγούν των ευθυνών του. Τώρα, η τρίτη πρόταση της Κομισιόν είναι να ζητηθεί από την πολιτική κατεύθυνση ε, για το αν δεν υπάρξει τελικά κάποια γνώμη από το Συμβούλιο. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και τι σε τι θα αντιστοιχούσε. Δεν ξέρω τι μιλάμε. Μιλάμε για μια νομική γνωμάτευση. Δεν έχω καταλάβει, σωστό όμολογο. Τέταρτη πρόταση και τελευταία θα ήταν να είναι δημόσια η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εφέσεων. Καλό είναι αυτό βέβαια πάντα, γιατί δίνονται κίνητρα κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και ε, αιτιολογούνται αποφάσεις. Αλλά δεν αρκεί να αιτιολογούνται οι αποφάσεις και η ψηφοφορία. Οι προτάσεις που σας κάνω εγώ είναι να βρούμε μια διέξοδο ε, από το έξοδο που βρίσκεται η Κομισιόν. Όταν τα κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει μια απόφαση, δεν μπορούν να λάβουν μια απόφαση. Άρα, το πρώτο που προτείνω είναι να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή συστηματικά να ακούμε από τα κράτη-μέλη τι αιτιολογία έχουν να προτείνουν. Να βγούμε από αυτήν ε, την αδιαφάνεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή γύρω από ε, τη διαδικασία της επιτροπολογίας που δεν ξέρουμε ποιος λέει τι, ποιος ψηφίζει τι και γιατί. Άρα αυτό το μέτρο θα ήταν πολύ σημαντικό. Δεύτερο, η εναλλακτική που προτιμώ και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο είναι στο πλαίσιο αυτών των εκτελεστικών πράξεων να κάνει κάποιε διακρίσει ανάλογα με τον τομέα, κάτι που υπάρχει ήδη. Για κάποιου τομεί που έχουν να κάνουν πραγματικά χάρη με την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και κάποια άλλα αισθήματα που θα πρέπει να οριστούν, που έχουν σημασία όμως για τους Ευρωπαίου πολίτες, φύση και τομέας για τα συγκεκριμένου αυτού τομεί να εξακολουθήσει να ισχύει ειδική πλειοψηφία. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αυτή την ειδική πλειοψηφία, τότε δεν δίνεται έγκριση. Δηλαδή έχουμε μια γενική εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης από τη στιγμή που δεν υπάρχει δική πλειοψηφία. Για κάποιους τομείς, για κάποια θέματα, για να μην μπλοκάρουμε βέβαια τη λειτουργία της Κομισιόν ούτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι οικολόγος, ε, αλλά δεν ε, το λέω αυτό ε, μόνο και μόνο για την οικολογία, γιατί έχουμε τα θέματα των τροφίμων, των μεταλλαγμένων και πολλών άλλων θεμάτων που άπτονται άμεσα της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρότεινα λοιπόν η Επιτροπή μας να προτείνει να γίνει διάκριση ανάλογα με τη φύση και τον τομέα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις άλλες εναλλακτικέ γιατί νομίζω ότι δημιουργούν περισσότερες αντιπαραθέσεις και σύγκρουση. Προσπαθώ λοιπόν να καταλήξω σε μια πρόταση για μια συνενετική διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το αδιέξοδο σε περίπτωση μη απόφασης από πλευράς ε, κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό. να διακρίνουμε το ουσιώδες από το περιτό. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και βέβαια με πολύ προσοχή θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δεν βλέπω κάποιον από τους σκιώδεις. Έχουμε για τους σοσιαλιστές το Ρίτσαλ, το Κόρμπε, το Μάικλ, για την Άλντε, αυτούς. Κάποιος που θα θέλει το λόγο. Ο Άσλι Φόξ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδη για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Δεν ξέρω, δεν το έχετε στι σημειώσει σα. Τέλο πάντων, ευχαριστώ παρόλα αυτά και ευχαριστώ και τον κύριο Ντύρα. Θέλω να πω ότι είναι πράγματι πρέπει να τροποποιηθεί αυτός ο τομέας νομοθεσία μεταξύ του 2011 και του 2015 36 40 υποθέσεις ε, που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Εφέσεων είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε γνωμοδότηση. Άρα φαίνεται ότι δεν αποδίδει αυτή η διαδικασία. Εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες η εξέταση, η διαδικασία της εξέτασης να γίνει πιο διαφανής ε, και σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση του κοινού στις ψηφοφορίες Επιτροπής Εφέσεων είμαστε υπέρ. Υπάρχουν και κάποιες επίμαχες βέβαια υποθέσεις. Εκεί το δικαίωμα θα, η Κομισιόν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ε, να παραπέμψει για γνωμοδότηση ε, την υπόθεση στο Συμβούλιο, ώστε να μπορούμε να δούμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις ε, μίας μία απόφασης. Μας ανησυχεί ως ομάδα ότι οι αλλαγές που προτείνουν τους κανόνες ψηφοφορίας της Επιτροπή Εφέσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Κομισιόν για να αποδυναμώσει τις εξουσίε των εκπροσώπων των κρατών μελό Και δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό η δική μου πολιτική ομάδα. Μας ανησυχεί επίσης το, η πρόταση ε, μείωση της απαρτίας στα 14 μέλη. Είναι πολύ χαμηλό αυτό το όριο. Θα συνεργαστούμε πάντως με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ή πρόεδρος, να υπενθυμίσω στους συντονιστές ότι το και οδό θα πρέπει να τα έχει η γραμματεία στη διάθεσή της, αλλιώς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ή ποια είναι η συντονίστρια και ο σκιώδης ε, ή ισκιώδης από την κάθε ομάδα. Δεν βλέπω συνάδελφο να θέλει το λόγο. Αυτή ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε τα πρώτα στοιχεία από τον εισηγητή μας. Στις 29 Μαΐου προβλέπεται να έχουμε την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης, η οποία θα σταλεί προς μετάφραση. Αυτό πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 10 Μαΐου, επομένως όποιος θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια κατηδίαν στον Πασκάλ Ντύρα, Α το κάνει πριν αυτή την ημερομηνία. Ο Πασκάλ επίση, αν θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με το εισηγητή από την Επιτροπή Γιούρη, χρήσιμο είναι αυτό πάντα, για να μην καταψηφιστεί ε, η γνωμοδότηση από μια άλλη επιτροπή. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, αν δεν θέλετε εσεί επίση το λόγο, μπορούμε να κλείσουμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό τη ημερήσια διάταξη. 12 Ιουλίου είναι η ψηφοφορία πριν το καλοκαίρι δηλαδή. Πριν πάνω στο 7, δύο ανακοινώσεις που δεν μπόρεσα να κάνω πριν. Η πρώτη είναι ότι οι συντονιστές συστήνουν να γίνει μια μεγάλη ακρόαση για το Brexit και τις συνταγματικές προκλήσεις και επιπτώσεις στις 20 Ιουνίου και όχι σήμερα. Αυτό βέβαια το είχαμε αποφασίσει ένα μήνα πριν, στην προηγούμενη συνδυασία. Και η δεύτερη απόφαση που έλαβαν οι συντονιστές ήταν ο Κρίστιαν Γιάν να είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης της έκθεσης ΠΕΤΗ για την νέα έκθεση Πυθαγένειας για το 2017. Αυτά. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7 της μερισιάς διάταξης που είναι νομοδότηση του κ. Ούλιας Ντόφσκι, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας Επιτροπής Γιούρη, για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015. Έχετε το λόγο κύριε Ουλιαντόσκη. Συνάδελφοι, πρόκειται για μια γνωμοδότηση που προσερτάται στην ε, ε, γνωμοδότηση της ε, Γιούρη που είναι η υπεύθυνη η αρμόδια από της Ουσίας Επιτροπή και αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Καταρχάς θα ήθελα να εστιάσω στην δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους θεσμούς και τα κράτη-μέλη αυτή είναι μια από τις, προ... απαιτήσεις που πρέπει να τηρήσουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την ε, κρίση ε, αλλά και για να επιτύχουμε την ε, σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εστιάσουμε σε διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα ορθολογισμός, εξοικονομήσεις όταν φτιάχνουμε νομοθεσία ώστε να μην δημιουργούμε νομοθετικό, νομοθετική υπερφόρτωση Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εφαρμογή σε, σε εθνικό επίπεδο είναι όταν οι οδηγίες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Όταν μιλάμε για την παρουσίαση όλων αυτών των νομοθετικών κειμένων στους πολίτες. Αυτά θα πρέπει να είναι διαφανή, γιατί αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη τους στην νομοθετική διαδικασία. Και έπειτα ο έλεγχος από τις ε, κοινή γνώμης όσον αφορά την εφαρμογή της κάθε νομοθεσίας στην πράξη να αναφέρω και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναφέρει ότι σε προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με την ε, νομοθεσία, την νομοθετική διαδικασία, το έχει ήδη αναφέρει, ε, δηλαδή το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εθνικών ε, κοινοβουλίων στην ε, ε, νομοπαραγωγική διαδικασία, το είπαμε και εχθές, και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι η εποπτεία όσον αφορά την εφαρμογή, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένα στοιχεία για το πώς προχωράει η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως λοιπόν θα πρέπει εδώ να δραστηριοποιηθεί περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Και νομίζω αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα που θέλησα να αναφέρω στη γνωμοδότησή μου και προσβλέπω στα δικά σας σχόλια και τις τροπολογίες σας. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ μικρή και μάλιστα έχουμε καθυστερήσει αν δούμε τις αρχικές προθεσμίες. Οπότε η Επιτροπή Γιούρι περιμένει τη δική μας απόφαση όσο γίνεται πιο σύντομα και αναφέρονται στο έγγραφό σας όλες οι σχετικές προθεσμίες. Αυτά λοιπόν και όπως σας είπα ε, περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, Κλαούντια Ταπαντέλα από τους Σοσιαλιστές είναι σκέδος για τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχουμε μία συγκεκριμένη θέση από πλευρά σοσιαλιστών, την οποία θα εκφράσουμε με τις ε, τροπολογίες που θα σας υποβάλλουμε. Πρώτα θα σας κάνω κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις. Ε, είμαι μέρος και της Επιτροπής Μεταφορών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και με λήψη μου διαπίστωσα από το 2016 κάποια κράτη-μέλη έχουν κάνει καταγγελίες για μάλλον έχουν ε, ε, ξεκινήσει διαδικασίε κατά κάποιων κρατών μελών ε, επί παραβάση, επειδή δεν έχουν μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν μια προσπάθεια για να επιταχύνουν την εφαρμογή των νομοθεσιών, αλλά και για να αποφύγουν την, την αμφισβήτηση του, του δικαίου. Έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Μπορούμε δηλαδή να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο των αποφάσεών μας. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν αυτές ε, ή να μην έχουν ε, στη ζωή των συμπολιτών μας. Αυτά έχω να σας πω και θα ε, υποβάλουμε τροπολογίες σε πιο λεπτομερείς. Ευχαριστώ πολύ. Oh, συγγνώμη ε, στο Μίχαλ Πόνεν, ο οποίο είναι ο σκιώδης για το ΕΛΚ. Μόλις το έμαθα. Ευχαριστώ πολύ ε, τον συνάδελφο για την συγκεκριμένη πρόταση και τι συστάσεις αναφορικά με αυτό εδώ το project. Συμφωνά με όλα όσα έχει παρουσιάσει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο σημείο 3 να τονίσουμε την σημασία της διαφάνειας και να κάνουμε και την ε, νομοθεσία ξεκάθαρη, κατανοητή και ακριβή. Στο σημείο 6 είναι πολύ σημαντικό στα εθνικά κοινοβούλια, αν έκανα κάποιες τροπολογίες, ε, νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξ αρχής. Όχι μόνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και σημαντικό είναι και το σημείο 10. για ε, τις διαδικασίες επί παραβάση και πριν την παράβαση. Δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη διαδικασία και σε αυτά. Υπάρχει μια η έκθεση λοιπόν της Γιούρη και σε αυτήν υπάρχουν στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του Ευρωπαϊκού Δικαίου το 2015. Γίνονται πολύ τυπικοποιημένα σχόλια σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες κτλ. Ξέρω ότι υπάρχουν πάνω από 100 τροπολογίες για αυτή την έκθεση. Ελπίζω σε συνεργασία με τη Γιούρη να καταφέρουμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την έκθεση, αυτή την πρόταση να επικεντρωθεί στο πραγματικό της πεδίο. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο σε εσά, γιατί δεν έχουμε άλλους σκιώδεις εδώ πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή και πάλι να σας ε, ενημερώσω όλους ότι με αυτή την έκθεση έπρεπε να διαπραγματευτούμε με τη Γιούρη να αναβάλουν την έγκριση της έκθεσης που ήθελαν να εγκριθεί ήδη τον Απρίλιο για να μπορεί η δική μας γνωμοδότηση να έχει ένα νόημα. Έγινε αυτό. Ε, ευχαριστώ για αυτή την παραχώρηση. Γι' αυτό πρέπει η τροπολογία σας να είναι στα αγγλικά, ώστε να ψηφίσουμε στις 29 Μαΐου και να είμαστε εντός της προθεσμίας ε, για τη διαδικασία. Σας ζητώ λοιπόν αυτό. Και τώρα ο λόγος πηγαίνει στον εισηγητή, αν θέλει. Ποια είναι η, η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 12 Μαΐου στις 6 μετά και μετά στις 29 θα γίνει εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία την ίδια μέρα. Οι τροπολογίες πρέπει να είναι στα αγγλικά. Τα ξεκαθαρίζω γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Εισηγητής, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ταπαρντάν και κύριε Μπόνη για τη γνώμη σας. Χαίρομαι που τα κέρια σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης ε, γίνονται αποδεκτά. Ξέρω ε, ότι καλό είναι να ενσωματώσουμε την άποψη όλων των ομάδων στο σχέδιο της νομοδότησης, γι' αυτό θα ήθελα να τα έχω γραπτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο, κλείνουμε αυτό το σημείο της σας διάταξης και πάμε στο τελευταίο, που είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, όλα τα τμήματα. Οι πολιτικές ομάδες τελικά αποφάσισαν ότι ε, αυτή η γνωμοδότηση που είχε γίνει παράδοση θα ε, δίνεται. Δεν είμαστε μία επιτροπή ε, που έχει να κάνει με τις δαπάνες, όμως έχουμε κάποιες ξεκάθαρες προτεραιότητες σχετικά με προγράμματα που θεωρούμε ότι έχουν επίπτωση στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και συνήθως η γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ έχει να κάνει με την αποφυγή περικοπών σε προγράμματα όπως Ευρώπη για τους πολίτες, ευρωπαϊκή εθαγένεια και άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την επικοινωνιακή τους πολιτική. Το 2019 θα έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις ευρωεκλογές. Η Κομισιόν ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τα κατάλληλα έγγραφα ε, που εξέδωσε και θεωρούμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τυχόν ανακοινώσεις, πληροφορίες και εκστρατείες που θα επέλθουν τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτά είναι και ο προϋπολογισμός του 2018 που τα χρηματοδοτεί. Αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή και όχι γνωμοδότηση για την εντολή ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τον τριμερή διάλογο στον κύριο Ζίγκριτ Μούρεσάν που είναι ο εισηγητής και της επιστολής αρχές Ιουνίου σχετικά με τις ε, τροπολογίες της ΑΦΚΟ στον προϋπολογισμό. Έχουμε στόχο να ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου, τη συνάντηση του Ιουλίου δηλαδή, επειδή δεν έχουμε άλλες συναντήσεις πριν την 31η Αυγούστου που είναι η προθεσμία φέτος για τις ε, ε, τροπολογίες των επιτροπών στη θέση του Συμβουλίου. Άρα, οι τροπολογίες θα βασιστούν στο σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής, ε, το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν και μετά ο εισηγητής θα το προσαρμόσει στις πιθανές αλλαγές που μπορεί να εισαγάγει το Συμβούλιο. Αυτή είναι λοιπόν η προσέγγιση. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον προπολογισμό τέλη Μαΐου. Θα στείλουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για μετάφραση στις 9 Ιουνίου. Και μετά θα γίνει η συζήτηση της γνωμοδότησης στις 20 Ιουνίου, όπως γίνεται και με την έκθεση του κυρίου Τιγιονοτόφσκη, θα είναι στα αγγλικά οι τροπολογίες. 22 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Αν κάποιος θέλει να δώσει κάποιες νέες ιδέες, ας το κάνει εγκαίρως. 12 Ιουλίου ψηφίζουμε στην ΑΦΚΟ, η τεχνική προσαρμογή στη θέση του Συμβουλίου μετά θα γίνει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αυτά είχα να πω. Χαίρομαι που συγκριτής εδώ. Έκανα μια εισαγωγή στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος ε, στην ΑΦΚΟ και τώρα, Ζίκφριτ, σου δίνω το λόγο για να μας πληροφορήσει σχετικά με το πώς θα γίνει η διαδικασία στην Επιτροπή προπολογισμού και πώς βλέπεις εσύ την όλη διαδικασία. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που με δεχτήκατε σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο επόμενο έτος. Τώρα είμαστε στα τελευταία στάδια. Το Μάρτι εγκρίναμε την έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές για το προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Εδώ σε αυτή τη φάση το Κοινοβούλιο λέει στην Επιτροπή στα δικά μας μάτια ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού την επόμενη χρονιά. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων θα καταθέσει το σχέδιο προϋπολογισμού η Κομισιόν στα τέλη Μαΐου και όπως ξέρετε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής θα ξεκινήσουν σε αυτή τη φάση. Στις κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν που εγκρίναμε το Μάρτι πρότεινα δύο βασικές προτεραιότητες. Νούμερο 1 Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας νούμερο 2, ασφάλεια των πολιτών, γιατί θεωρώ ότι αυτό περιμένουν από την Ένωση οι πολίτες αυτή τη στιγμή, δουλειές και ασφάλεια. Και πώς θεωρώ ότι θα το πετύχουμε αυτό. Πρώτον, για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας χρειαζόμαστε μια ισχυρή ανταγωνιστική αξιόπιστη οικονομία που θα την εμπιστεύονται οι επενδυτές και ο ιδιωτικό τομέας. Και γι' αυτό θα ήθελα να εφαρμόσουμε τα προγράμματα τα οποία επενδύουν χρήματα στις υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των επιχειρηματιών, κυρίως των νέων και την ανεργία των νέων. Τα προγράμματα λοιπόν που προτείναμε να εφαρμοστούν είναι ο ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, κόσμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εράσμους. Ε, όχι μόνο ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, βελτιώνει τις ε, πιθανότητες στην αγορά εργασίας, γιατί σήμερα στην Ευρώπη πάνω από 60% των εργοδοτών θα δώσουν τη δουλειά σε ένα νέο που έχει διεθνή εμπειρία. Και φυσικά η απασχόληση για τους νέους, η πρωτοβουλία αυτή. Υποστηρίζω την προπαρασκευαστική ε, δράση ε, ενώπιον της πρότασης της Κομισιόν ε, γιατί τα δημόσια κονδύλια είναι λίγα και το να δίνεις χρήματα σε 28 κράτη-μέλη για πράγματα τα οποία μεμονωμένα θα δώσουν ίδια αποτελέσματα δεν είναι τόσο σόφρον, είναι καλύτερο να δώσεις τα χρήματα σε νοσιακό επίπεδο. Τώρα, για την και τώρα για το γεγονός ε, ότι στο παράρτημα 3 και 4 έχουμε περιορισμένους πόρους, ε, πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε κάτι με τους περιορισμένους αυτούς πόρους τα γραφεία οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, Europol, just front, εξτεάζω θέλουν να αυξήσουν το προσωπικό τους για να προστατέψουν καλύτερα τα εξωτερικά σύνορά μας, να έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών σχετικά με τους ε, τομείς της τρομοκρατίας, ε, της, ε, του λαθρεμπορίου όπλων και ανθρωπίνων όντων ε, για να ε, δούμε και το θέμα της άμεσης γειτονίας μας, ε, της ανατολικής γειτονίας που αντιμετωπίζει μια ρωσική ομοσπονδία όλο και πιο ενεργή και της νότιας γειτονίας όπου έχουμε πολλές προκλήσεις λόγω των προσφύγων και της μετανάστευσης, ακόμα και παράνομης μετανάστευσης. Πέρυσι, κάναμε μια αποστολή στο Λίβανο με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και είδαμε ότι είναι πιο εύκολο και πιο ασφαλές να έχουμε ε, τους πρόσφυγες εκεί. Γιατί εκεί στοιχίζει 1.000 ευρώ το χρόνο για να τους ε, διαχειριστείς, ενώ στην Ένωση 6.000, πολλές φορές και παραπάνω. Όταν ε, τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να επιστρέψουν. Άρα είναι καλό να τους κρατήσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη χώρα προέλευσης. Αυτές πρέπει να είναι οι μεγάλες προτεραιότητες. Να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα. Ειδικά τώρα που ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσες ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Οι κατάλληλοι πόροι ε, για τις αντιπροσωπείες ε, της Κομισιόν, για τον διάλογο με τους πολίτες, ε, για διάφορες δράσεις εταιρικέ, όλα αυτά είναι επίσης σημαντικά. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι συμφωνήσαμε στο 7 πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Το 2014 ε, πολλές από τις προκλήσεις που έχουμε σήμερα όπως η έλλειψη ασφάλειας, η τρομοκρατία, η μετανάστευση δεν ήταν προβλέψιμες και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Η διαδικασία ξεκίνησε, εμείς συμφωνήσαμε επί του πακέτου με το Συμβούλιο, εμείς στο Κοινοβούλιο όμως κάναμε τη δική μας δουλειά. Σωστά, το εγκρίναμε πολύ γρήγορα, τώρα θα εγκριθεί, ε, ε, υποτίθεται ότι θα εγκρινόταν ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της περισμένης εβδομάδας, όμως το Ηνωμένο Βασίλειο δυστυχώς είπε ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα μπορέσουν να το υποστηρίξουν. Άρα η αναβολή δύο-τριών μηνών ε, μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι μετά τις εκλογές δεν είναι μεγάλο ε, πρόβλημα, αλλά το να μην γίνει η αναθεώρηση η οποία θα αυξήσει τα ταβάνια, την, ε, το ανώτατο όριο 1,5 δις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις δράσεις που θέλουμε Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε, 200 εκατομμύρια, 1,2 δις για την ανεργία. Όλα αυτά, αν δεν γίνουν, μέσω της αναθεώρησης θα είναι πολύ δύσκολο του χρόνου να έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος ε, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε το 2014. αναβολη 2 2-3 μηνών είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, είναι κατανοητό λόγω των εκλογών στο ΕΒ Βασίλειο, όμως τελικά πρέπει να γίνει η αναθεώρηση και πρέπει να πω ότι 200 εκατομμύρια πάνε στην έρευνα και στην καινοτομία. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος ε, ωφελούμενος από τον ορίζοντα 2020 είναι το Ηνωμένο Βασίλειο το 2016. Γιατί, γιατί τα πανεπιστήμια τους πηγαίνουν παντού στον κόσμο, έχουν εξαιρετική έρευνα. Είναι ο βασικός ωφελούμενος λοιπόν και, είναι και θέλουν να υπάρξει αυτή η αύξηση των κονδυλίων. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε από τη δική μου πλευρά σχετικά με το που βρίσκεται τώρα ο προϋπολογισμός. Θέλω η παρουσία μου σήμερα εδώ να είναι η αρχή της συνεργασίας μας για αυτό το έτος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να γνωρίζω ότι αφότου η Επιτροπή δημοσιεύσει τη δική της θέση θα μπορέσουμε εμείς να μείνουμε σε επαφή μέχρι τα τέλη ε, της διαδικασίας ε, για να μπορέσω να λάβω υπόψη τις ανησυχίες σας στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Περιμένω λοιπόν τη γνωμοδότησή σας τώρα για τους τομείς που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση το επόμενο έτος μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης. Όπως ξέρετε, για τα πιλωτικά project, τα μέλη της, Επι... Επιτροπή οι πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές ε, μπορούν να κάνουν τέτοια πιλωτικά ε, έργα και η δική σας Επιτροπή το έχει κάνει πολλές ε, έτσι πρέπει λοιπόν να στείλετε μέχρι σήμερα το μεσημέρι όλα τα πιλωτικά προγράμματα που θέλετε, στα οποία θέλετε να συμμετάσχετε σε εμά. Εμείς θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε ε, αυτό το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να κάνει ένα πακέτο που θα προτείνει χρηματοδότηση για τα πιλωτικά project ε, όπως έγινε και πέρυσι. Εγώ ήθελα ένα τέτοιο project, το κατέθεσα, πήγε στην προαξιολόγηση. Από αυτή την άποψη λοιπόν αδειμονώ για τη συζήτηση μαζί σας και για την γνωμοδότηση της Επιτροπής σας. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι εσείς ε, τη συντάσσετε και θα την καταθέσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την εισαγωγή. Ο κύριος Ιασδόσκη νομίζω ότι ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, ιδίως ε, σε σχέση και με, τη, με το σχέδιο του υπερπολογισμού επί το οποίο και εργαζόμαστε. Μιλάμε για το σχέδιο προπολογισμού για το 2018. Έχω κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσον ήδη από τώρα μπορούμε να συζητήσουμε τόσο αναλυτικά τον προπολογισμό στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ωστόσο, Οφείλω να πω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω τον κατάλογο προτεραιοτήτων σας, μετανάστευση, ανατολική εταιρική σχέση, ιδίω όλοι αυτοί οι τομείς. Είναι τομείς στους οποίους η Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Εμείς όμως ως Επιτροπή ΑΦΚΟ θα έπρεπε ίσως να εστιάσουμε σε κάτι άλλο. Ως Επιτροπή ΑΦΚΟ θα έπρεπε να φροντίσουμε ορισμένες διατάξεις ε, του, της συνθήκης για τον προλογισμό να εφαρμόζονται, να τηρούνται. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, να ε, ελέγχουμε τη συμμόρφωση των διατάξεων του προπολογισμού σε σχέση και με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, την εποπτεία και τη ενέργεια ελέγχων. Ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον τελικά εφαρμόζονται οι κανόνες του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Ίσως μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό από κοινού. Η πρόεδρος δεν βλέπω κάποιον να θέλει το λόγο. Το έχω ξαναπεί. Ίσως όμως καλό θα ήταν να επαναλάβω κάποια από τα σχόλια που έκανα πριν παρουσία του κυρίου Μουρεσάν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμάς στην ΑΦΚΟ. Κάποια θέματα που αφορούν την ουσία να ληφθούν υπόψη. Όπως γνωρίζετε, γιατί αναφέρατε και εσείς ο ίδιος τη σημασία της επικοινωνίας με τους πολίτες. Δεν είμαστε τα πανάρα, δεν έχουμε πρόβλημα ε, ως προς αυτό. Αλλά το 2018 θα είναι ένα έτος που βλέπω ήδη ότι η επικοινωνία σε σχέση και με την ευαισθητοποίηση για τις ευρωεκλογές του 2019 θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μετά τη Λευκή Βίβλο, ήδη από φέτος νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις ε, εκστρατείες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, ώστε να συμμετέχει πλώς πολίτης στις συζητήσεις. Δέχομαι τι προτεραιότητές σας, ε, είναι θεμελιώδης για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, πιστεύετε όμως επίσης ότι ο προπολογισμό αυτός θα πρέπει να είναι αρκετά σημαντικός ό,τι αφορά την ε, επένδυση στην επικοινωνία. Άρα ελπίζω στο πρόγραμμα ε, για τους πολίτες και στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους πολίτες να μην υπάρξουν περικοπές και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες ε, επικοινωνίας που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές και είναι καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμών και όχι μόνο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και όλων των θεσμικών οργάνων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και θα έχουμε πολλές, ε, έχουμε πολλές προσδοκίες και από τις δράσεις που θα οργανωθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Θα προετοιμάσουμε αντί για γνωμοδότηση μια επιστολή που θα σας τη στείλουμε σε ό,τι αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει αρχές Ιουνίου ε, εφόσον θα έχουμε δει και την πρόταση της Κομισιόν. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, τροπολογίες, γιατί έπεται και το καλοκαίρι και υπάρχει λιγότερη ευελιξία για συναντήσεις με την Κομισιόν. Θα καταρτήσουμε τροπολογίες, θα τις ψηφίσουμε τον Ιούλιο και επίσης ε, προσπαθήσουμε να έχουμε επαφή με τον εισηγητή για να γίνει μια προσαρμογή όταν θα ξέρουμε ε, τι θα γίνει και με την Κομισιόν, ε, συγγνώμη, το Συμβούλιο, γιατί προς αυτούς θα απευθύνουν τροπολογίες μας. Ελπίζω αυτό να μην είναι πρόβλημα και για σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε πάρα πολύ. και σε ό,τι αφορά τα τέσσερα πιλωτικά. Είχαμε τις εστάσεις των ε, συντονιστών. Ελπίζουμε να είναι γενναιόδορη κομισιόν τη Δεν έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα. δεν είναι στο δικό σα ε, χέρι, για δεν ασκώ πιέσει ε, σε εσά. ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από ό,τι βλέπω. Ζίγκριτ, θες να μιλήσεις. Αν όχι, σε ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ ολοκληρώσαμε, που σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας. Αλλά έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι, παρουσία του κυρίου Τίμερμανς. Πολιτική Σύμβουλη, συνεργάτες, παρακαλώ, ενημερώστε τους βουλευτές σας για την έκτακτη συνεδρίαση και στις συντονιστές τα συζητήσαμε ε, τι θα κάνουμε για να κάνουμε δύσκολη τη ζωή του κύριου Τίμπερμαν ε, στην ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ.